Bom dia, vamos Καλημέρα σας. Ας αρχίσουμε με τις εργασίες μας. Temos para Για να αρχίσουμε λοιπόν, προβλέπετε μια συζήτηση ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα, μια εμπορική ανισορροπία θα πρέπει να λήξει η συζήτηση κατά τις 9.30 για να αρχίσουμε με τις ψηφοφορίες. Θα ήθελα να έχετε την κάρτα σας ε, μαζί, εάν χρειαστεί, γιατί μπορεί να χρειαστεί. Για το, δεύτερο, για το πρώτο αυτό θέμα λοιπόν, ο κύριος Στέρξ έχει το λόγο από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι οι σχέσεις μας με την Κίνα είναι πολύ σημαντικές. Δεν πρέπει να τις κοιτάμε ελαφρά την καρδία. Έχω περιορίσει βέβαια τα θέματα που περιλαμβάνω γιατί είναι κάποια θέματα που πρέπει να σκεφτεί δικιά μας η Επιτροπή και αυτό είναι κυρίως οι κοινωνικές πτυχές των ε, εμπορικών σχέσεών μας με την Κίνα. Υπάρχει έτσι κι ένα ερωτηματικό στον τίτλο της γνωμοδότησης. Υπάρχει ή δεν υπάρχει εμπορική ανισορροπία στις ε, σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα. Αυτό πρέπει να δούμε. Υπάρχουν ε, κάποια στοιχεία ανισορροπίας πράγματι αλλά στη συζήτηση πρέπει να μπούμε πολύ σε βάθος για να τα βρούμε και να μην ε, κοιτάμε επιφανειακά το θέμα. Από τις σχέσεις μας, τις εμπορικές με την Κίνα, έχει πέσει το ισοζύγιο, το δικό μας το εμπορικό η επιτυχία της Κίνας είναι μεγάλη όσον αφορά τις επενδύσεις στις, στις δικές μας χώρες. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό και να το υπογραμμίσουμε. Είναι επίσης προφανές ότι η Κίνα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εμπορικούς εταίρους διεθνώς και το γεγονός ότι εδώ και κάποια κάπου 10 χρόνια περίπου έχει μια ανοιχτή οικονομία και αποτελεί μέρος της παγκόσμιας οικονομίας πια, αυτό δημιουργεί και κάποιες υποχρεώσεις στην Κίνα. Η, την Κίνα λοιπόν πρέπει να τη δούμε διαφορετικά σήμερα από ό,τι τη βλέπαμε πριν από 10 χρόνια. Έχουμε κάθε συμφέρον να συζητάμε με τους Κινέζους για τα κοινωνικά ζητήματα και τις κοινωνικές προδιαγραφές. Το λέω και στην γνωμοδότησή μου ότι πρέπει να δούμε τα θέματα τα κοινωνικά όχι μόνο με την Κίνα, γιατί σε ολόκληρη την Ασία υπάρχουν ε, χώρες με τις οποίες πρέπει να συζητήσουμε για τα κοινωνικά θέματα. Αναπτύσσεται η Κίνα και υπάρχουν επιχειρήσεις λοιπόν που φεύγουν από την Κίνα και πηγαίνουν και καθίστανται σε άλλες ασιατικές χώρες. Οπότε και εκεί πρέπει να δούμε τι κοινωνικές ηθίκες επικρατούν σε αυτές τις επιχειρήσεις που καθίστανται σε άλλες χώρες. Στην Κίνα βέβαια βλέπουν τα πράγματα κάπως διαφορετικά από ό,τι τα βλέπουμε εμείς πολλές φορές. Αυτό ισχύει για την κοινωνική πολιτική, για την κοινωνική ασφάλιση. Οι προδιαγραφές είναι διαφορετικές εδώ από ό,τι στην Κίνα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν υπάρξει πολύ σημαντικές εξελίξεις στα κοινωνικά ζητήματα. Υπάρχει νομοθεσία για τα εργασιακά που έχει φτιαχτεί από ειδικού της δικιάς μας Υπήρου και η κινέζικη κυβέρνηση έτσι λοιπόν κοιτάζει με ιδιαίτερη προσοχή πώς εμείς διευθετούμε τα κοινωνικά ζητήματα στις χώρες μας. Είναι προφανές λοιπόν ότι εφόσον η Κίνα θέλει να αποτελέσει μέρος της παγκόσμιας εμπορικής κοινότητας πρέπει να ακολουθεί και τους διεθνείς κανόνες εμπορίου. Και εκεί είναι που αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Και γι' αυτό και η γνωμοδότησή μου μιλάει για ελεύθερα συνδικάτα, και μιλάει όχι μόνο για την ύπαρξη νομοθεσίας αλλά και για την εφαρμογή και τον έλεγχο της νομοθεσίας αυτής. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη δηλαδή. Είναι συνεπώς πολύ σημαντικό οι Κινέζοι να ασχοληθούν με την ανάπτυξη κοινωνικής νομοθεσίας και νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης, να μην υπάρχουν ανισορροπίες στην αγορά και είναι προφανές ότι οι Κινέζοι πολίτες αποταμιεύουν πολύ λιγότερα για τις συντάξεις τους ατομικά. Βασικά υπάρχει μεγάλη ανισορροπία ανάμεσα στην εσωτερική κατανάλωση και στις εξαγωγές. Δηλαδή ατομικά δεν τα πανάνε πολλά χρήματα οι Κινέζοι. Η ανάπτυξη βέβαια είναι 7%, δεν είναι 10-11%. Και ο εσωτερικός πλούτος είναι της τάξης του 7%. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρυνθεί η εσωτερική κατανάλωση επίσης. Συμβαίνουν αρκετά πράγματα βέβαια τα τελευταία χρόνια που δεν συνέβαιναν παλιότερα. Συνεπώς κύριε Πρόεδρε, πιστεύω και επίτηδε, δεν έχω κάνει μια μεγάλη γνωμοδότηση. Πιστεύω πάντως ότι η γνωμοδότησή μου περιλαμβάνει κάποια από τα πιο σημαντικά ζητήματα. Και έτσι μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς στη συζήτηση που γίνεται στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Επαναλαμβάνω ότι οι σχέσεις μας, οι εμπορικές σχέσεις μας με την Κίνα είναι κάτι πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να το βλέπουμε περιθωριακά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την εισήγηση αυτή. Νομίζω ότι ήδη θίξατε ορισμένα βασικά θέματα, σημαντικά θέματα, που πλαισιώνουν αυτή τη γνώμη και θα απασχολήσουν και την Επιτροπή μας. Και θα απασχολήσουν και την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Πλάμ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω όλους τους συναδέλφους και ιδίως τον εισηγητή. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια και θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή ιδιαίτερα για την παρουσίαση που έχει κάνει και νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι ιδέες που υπογράμισε. Εγώ θα ήθελα να μου επιτρέψετε να θίξω ορισμένα ζητήματα τα οποία για μένα είναι ουσιώδη. Οι Κινέζοι είναι από τους πιο σημαντικούς παίκτες μέσα σε εισαγωγικά σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας στα πλαίσια μιας συμφωνίας ε, εταιρικής σχέσης και σύνδεσης ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο το εμπόριο μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωση. Θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι, ξεκινώντα από αυτά που είπε ο, ο εισηγητής, δηλαδή την ανάγκη για κοινωνικό διάλογο, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα χαρακτήρα ηγετικό σε ό,τι αφορά τις εργασιακές συνθήκες και την αντιμετώπιση των εργασιακών και κοινωνικών θεμάτων σε παγκόσμιο κόσμο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε κοινωνικού χαρακτήρα συμφωνίε και συμμαχίε με αυτόν τον παγκόσμιο παίκτη που είναι η Κίνα. Δηλαδή να υπάρξουν κοινέ αντιμετωπίσει στα κοινωνικά θέματα μεταξύ ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα, ώστε να έχουμε κοινά εργασιακά πρότυπα τα οποία θα ανταποκρίνονται σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ στην ε, ρήτρα εταιρική υπευθυνότητα σε ό,τι αφορά τα θέματα των επενδύσεων που γίνονται στην Κίνα. Πιστεύω ότι οι επιχείρησεις αυτές μπορούν να διαδραματίσουν ένα μεγάλο ε, ένα σημαντικό ρόλο για να προωθήσουν την ε, εδραίωση προτύπων στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο λοιπόν θα πρέπει να εστιάσουμε, να δώσουμε έμφαση στην κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. και να εξασφαλίσουμε ότι η προστασία των εργαζομένων και η γενική κοινωνική προστασία θα πρέπει να υπογραμμιστούν επίσης. Το 2006 ήδη η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των, του ΟΗΕ τόνισε την ανάγκη να γίνεται κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες η εργασία, ιδίως σε ό,τι αφορά τα ρελέ. Και επίσης τόνισε και πρέπει να τονίσουμε επίσης τη σημασία της βοήθειας που δίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αναπτυξιακών εργαλείων σε τρίτες χώρες. Θα πρέπει επομένως να υπάρξει μια συμμαχία με την Κίνα για την βελτίωση της εκπαίδευσης κατάρτισης, την εκρίζωση της ένδυας, τις καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας. <clears throat> για όλους αυτούς τους λόγους είναι απαραίτητη μια καλύτερη συνεργασία με την Κίνα για να υπάρξει καλύτερη προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και των μεταναστών εργαζομένων, μια μέρημνα για την ισότητα ευκαιριών για τα δύο φύλλα και η μεταλαμπάδευση βελτίστων πρακτικών σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε την ε, δυνατότητα συνεργασίας για τη δημιουργία πρασίνων θέσεων εργασίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε τις νέες κλιματικές και ενεργειακές προκλήσεις. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά στοιχεία που θα ήθελα να υπογραμμίσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χέλμερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι συνειρπασμένος από αυτά που ακούω. Πόσοι από εσά άραγε έχετε μπει σε ένα θάλαμο, σε ένα υπνοτήριο μάλλον εργαζομένο σε κινέζικα εργοστάσια για να δείτε σε τι συνθήκες ζουν αυτοί οι άνθρωποι, ποια είναι η πραγματικότητα της εργασίας και της διαβίωσής της. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον κύριο Στέρξ και θέλω να τον ευχαριστήσω για το πολύ καλό έργο το οποίο έχει φέρει σε πέρας, αλλά έχω κάποιες ε, αμφιβολίες για τον αντίκτυπο του έργου του σε πραγματικό επίπεδο. Μιλάμε για το εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνα. Η Κίνα έχει κάνει μια τεράστια συμβολή στη μείωση του πληθωρισμού στην Ευρώπη με το να κάνει διαθέσιμα αγαθά σε προσβάσιμες τιμές. Αλλά θα πρέπει να ανησυχήσουμε λιγάκι γιατί αυτή η εποχή έχει πλέον παρέλθει. Οι Κινέζοι εργαζόμενοι έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, να πληρώνονται περισσότερο και αυτή είναι η στόχη στους οποίους εμείς θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Να υπενθυμίσω όμως συναδέλφους ότι υπάρχει ο σιδηρούς νόμος της οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης ότι τα πρότυπα εργασίας και οι συνθήκες εργασίας αλλά και του περιβάλλοντος επί τη ευκαιρία βελτιώνονται όταν μια, κοινότητα, μια οικονομία περνάει ένα κατόφλι ευμάρειας. Βλέπουμε τώρα να γίνεται αυτό στην Κίνα, να υπάρχει πίεση για αύξηση των αποδοχών. Πολλές επιχειρήσεις πληρώνουν υψηλότερες αποδοχές. Αυτό είναι όλα, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα υποστηρίζαμε εμείς. Αλλά όλα αυτά καθοδηγούνται από μια γενική οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη στη χώρα αυτή. Και εμείς τώρα το να είμαστε εδώ και να κηρύττουμε από καθέδρα σε σχέση με αυτά τα οποία γίνονται στην Κίνα, αυτό δεν έχει νόημα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλέ σοβαρέ παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Υπάρχουν άτομα τα οποία συλλαμβάνονται στι 3 η ώρα το πρωί, και του πηγαίνουν σε στρατόπεδα κατουμένων και βασανίζονται. Η Κίνα είναι πάρα πολύ διστακτική να συζητήσει τέτοιου είδου θέματα ή να ανταποκριθεί στην πίεση τη δύση για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά τα θέματα θα πρέπει να είναι εκεί που εστιάζουμε την προσοχή μα. Αν τώρα θεωρείτε ότι εμείς θα πρέπει να κάνουμε ε, αιτήσει προς την Κίνα για καλές συνδίκες εργασίας ή ισότητα των φίλων στην Κίνα, αυτό είναι χάσιμο χρόνο. Και εδώ ουσιαστικά αντιδρούμε σε μια έκθεση η οποία ακόμα δεν έχει διατυπωθεί πλήρως σε έγγραφη μορφή. Και είναι υπερβολικό ίσω να έχουμε μια γνωμοδότηση για μια έκθεση η οποία δεν έχει ακόμα περατωθεί. Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε αυτή την ευκαιρία για να δείξουμε ότι έχουμε κοινωνική ευαισθησία και συμπάθεια και κατανόηση για τους εργαζομένους σε μια μακρινή χώρα, αλλά κανείς στην ε, Κίνα δεν θα δώσει διάραμα μάλλον για όλο αυτό το θέμα. Αυτό ήθελα να πω εξ όνομα της ομάδας μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χέλμερ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάν. Μπορούμε βέβαια να σταυρώσουμε τα χέρια και να μην κάνουμε απολύτως τίποτα για τα θέματα αυτά. Να πούμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται, αλλά να μην κάνουμε τίποτα. Να κάνουμε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα έγινε κάτι τέτοιο σε ό,τι αφορά την κλοπή της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς των ε, ε και της καταπίεσης που αντιμετωπίζουν από την Κίνα. Λοιπόν, δεν αρκεί να κατονομάσουμε τα γεγονότα, αλλά νομίζω ότι η, ε, η αντιμετώπιση είναι σωστή αυτή που ανεφέρθηκε, ότι τι κάνει μια γιγάντια χώρα όταν του λένε, της λένε οι άλλοι τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να λάβουμε υπόψη πολύ σωστά την πολιτική διάσταση, όπως έκανε ο κύριος Στέρξ. Πρέπει η στάση μας να είναι join the game, να μπορέσουμε να έρθουμε σε επίπεδο να βοηθήσουμε τους Κινέζους να είναι μέσα στο παγκόσμιο παιχνίδι. Γιατί παραδείγματο χάρη όταν γίνουν μέλη του ΠΟΕ θα πρέπει να παίζουν και με του κανόνε του ΠΟΕ. Η πίεση πρέπει να παραμείνει προ την κατεύθυνση τη Κίνα. Αλλιώ θα αφήσουμε την Κίνα να κάνει ό,τι θέλει, να αντιμετωπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά το αδοκούν. Πρέπει επομένω να παραμείνει μια πίεση προ την Κίνα από την διεθνή κοινότητα γιατί όπω ελέγχθη πράγματι έχουν πετύχει κάτι οι εργαζόμενοι στην Κίνα, έχουν περισσότερα χρήματα, έχουν περισσότερη ελευθερία, έχουν γίνει πολλά πράγματα τα οποία στο παρελθόν δεν ισχύαν. Αλλά <clears throat> δεν είναι επαρκή αυτή η πρόοδος. Γι' αυτό πιστεύω κύριε Στέρξ θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να θέσουμε περαιτέρω απαιτήσει, να μην θεωρήσουμε ότι έχουν τελειώσει όλα αυτά τα προβλήματα. Παραδείγματο χάρη στον τομέα τη ε, κλωστοφαντουργία. Σε πολλέ περιοχές της Κίνας που έχει συμφωνίες με τις ε, κλωστοεφαντουργικές βιομηχανίες της ε, Ευρώπης θα πρέπει να τηρηθούν οι κανόνες οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί. Δεν πρέπει λοιπόν αυτά τα οποία κάνουμε να είναι μια σταγόν εν το ωκεανό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει πρόοδος στα θέματα αυτά. Κάτι ακόμα Εμεί υποστηρίζουμε τις δομές ενός συστήματος κοινωνικής οικονομίας τη αγορά. Αυτό συμπεριλαμβάνει και την υπευθυνότητα των επιχειρήσεων. <clears throat> Θα έπρεπε λοιπόν οι Κινέζοι να ανταποκριθούν στην απέτηση για ένα τέτοιο σύστημα. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να φτάσει στο σημείο μια συμμαχία στα κοινωνικά θέματα, αλλά τουλάχιστον μια προσέγγιση. Παραδείγματο χάρη να μην υπάρχει η παιδική εργασία η οποία υπάρχει. Και τώρα βρισκόμαστε εξάλλου σε μια εποχή γενικού αλφαβητισμού σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρονικά θέματα. Σε μια εποχή που υπάρχει παγκόσμια γνώση και παγκόσμιο ίντερνετ θα πρέπει η γνώση να φτάσει όλους και στην Κίνα και εκείνα να κάνει ό,τι είναι δυνατό ώστε να μπορούν τα άτομα να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, να δουν τι μπορούν να αναλάβουν από το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και τι δεν μπορούν να, ή δεν θέλουν να αναλάβουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στους τομείς της Ασφάλεια και τη υγεία στην εργασία. Μια τέτοια λοιπόν πρωτοβουλία θα ήταν πάρα πολύ θετική για του εργαζόμενους και στην Κίνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος. Άλλοι τρει έχουν να λάβουν το λόγο. Θα ήθελα να σα ζητήσω να μην μακρηγορείτε και να περιοριστείτε στα ουσιώδη, ώστε να περάσουμε στη συνέχεια στην ψηφοφορία. Θα δώσω λοιπόν το λόγο

πω ότι η Κίνα είναι 200, 200 χρόνια μπροστά. Εμείς ανεβαίναμε στα δέντρα όταν η Κίνα είχε ένα οργανωμένο κράτος και μπορούμε να εγκρίνουμε όσα ψηφίσματα θέλουμε, αλλά όταν ο Κινέζος ε, πρόεδρος έρθει στη Γαλλία και παραγγείλει 200 Airbus, τότε όλα έχουν καλώς. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είμαστε πια τόσο υποκριτές ε, στην προσέγγισή μας. Ξέρω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατώνται στην Κίνα. Ξέρω ότι δεν μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν στα συνδικάτα. Αλλά όσο αναπτύσσεται η μεσαία τάξη στην Κίνα, η Κίνα, η τάξη αυτή θα λάβει αυτά που υπάρχουν πλέον, είναι δεδομένα στην Κορέα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και εκεί κάποτε ήταν δικτατορία. Και νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις αλλαγές που θα πρέπει να επέλθουν στην Κίνα. Αλλά όταν βρεθείτε στο αεροδρόμιο των Βρυξελών, έχουμε σωρία προϊόντων τα οποία κατασκευάζονται στην Κίνα. Κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη διότι πολλά προελέχθησαν. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Στέρξ και σε μια πολύ σύντομη έκθεση έθιξε σωρία θεμάτων. Δεν αναφέρθηκε μόνο στην Κίνα αλλά και σε άλλες ασιατικές χώρες που αναφέρθηκαν στο σημείο 5. Συμφωνώ με τον Τόμας Μαν, είναι σταγόνα εν το ωκεανό. Και είναι πολύ απογοητευτικό όταν λέμε, λέμε, λέμε και δεν γίνεται τίποτα. Το ίδιο νιώθουμε όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι σαν να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο αν μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Αλλά θα πρέπει να έχουμε ενιαία φωνή με τις ΗΠΑ γιατί μιλάμε για ένα δις ανθρώπων που είναι εμπορικοί εταίροι της Κίνας και θα πρέπει να ορίσουμε συγκεκριμένους όρους όταν μιλάμε για μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και συμφωνίες. Η κατάσταση δεν είναι τόσο καλή όσο θα μπορούσε, θα πρέπει να επέλθουν ε, βελτιώσεις και αυτό θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Η κυρία Κρίστες, ο κύριος Er- Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βεβαίως, η Κίνα είναι εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματικός εμπορικός εταίρος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προβάλλουμε απαιτήσει, διότι δεν υπάρχει τήρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Γίνονται σοβαρές παραβιάσεις. Στην Αγγόλα το 2009 είχαμε διαπιστώσει ότι κατά την ε, κατασκευή ε, ε, ενός γηπέδου για το πρωτάθλημα της Αφρικής, τότε ε, οι εργαζόμενοι ήταν Κινέζοι και μόνο κινέζικα υλικά είχαν χρησιμοποιηθεί δεν υπήρχε ούτε ένας Αφρικανός ε, εργάτης επιτόπου. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να δεχτούμε Δεν μπορούμε να δεχτούμε να μην γίνονται αυτές οι εργασίες υπέρ των Αφρικανών και βεβαίως και η απόφαση των Κινέζων και ως προς το, ως προς το θέμα κατά πόσο οι κατάδικοι έπρεπε να μείνουν στις φυλακές ή να ε, εργαστούν, είχαμε κρίνει, είχε κρυφθεί τότε ότι καλύτερα πρέπει, θα ήταν να εργαστούν. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο ο συνάδελφος Στέρξ θέλει να σχολιάσει. Μπορεί, εντάχει. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα και με τον κύριο Χέλμετ ότι δηλαδή η βελτίωση των κοινωνικών προδιαγραφών συνάδει με την ευημερία, πάνε χέρι-χέρι. Αν έχουμε καλύτερες συνθήκες στην κοινωνία, ε, υπάρχουν εξελίξεις και στις κοινωνικές προδιαγραφές. Τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε δει θεαματικές αλλαγές στην Κίνα. Συμβαίνουν πολλά πράγματα εκεί. Μπορεί να μην είναι αρκετά καλά για τις δικές μας τις προδιαγραφές, αλλά αν συγκρίνεται την κατάσταση ε, σήμερα ε, με τους ανθρώπους που φεύγουν από την Ήπεθρο και πηγαίνουν στα αστικά κέντρα, διαπιστώνουμε ότι βελτιώνεται σημαντικά το επίπεδο ζωής τους. Υπάρχει τεράστια βελτίωση επίσης σε σύγκριση με τι συνέβαινε εκεί πριν από 30 χρόνια. Άρα εξέλιξη προς το καλύτερο υπάρχει. Δεν συμφωνώ μαζί με τον κύριο Χέλμετος προς το Ότι μένουμε, ότι μάλλον πηγαίνουμε προς τα πίσω αντί να πηγαίνουμε προς τα μπρος. Όχι. Και δεν είναι αλήθεια ότι οι Κινέζοι δεν μας ακούνε. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας πάντα ότι στο εσωτερικό της Κίνας, για τα ίδια αυτά θέματα, για την κοινωνική οργάνωση δηλαδή λοιπά υπάρχουν συζητήσεις που γίνονται και σε ηγετικό επίπεδο. Σίγουρα είναι δύσκολο, είναι ένα πάζλ, είναι δύσκολο να πούμε ότι ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, δεν είναι η δημοκρατία η ανοιχτή που όλα γίνονται γνωστά ε, στη δημόσια σκηνή, όχι. Αλλά έχουμε συζητήσει πολλές φορές με την κινέζικη αντιπροσωπεία για αυτά τα θέματα και ο Στίβεν Χιούζ, ο συνάδελφός μας, ο σοσιαλιστής, όταν ε, συζητάμε για την ασφάλεια στα ορυχεία, να ξέρετε ότι έχει δουλέψει χρόνια και χρόνια για να υπογραφεί ένα πρωτόκολλο το οποίο θα βελτιώνει την ε, κατάσταση ασφάλειας στα ορυχεία και μπορεί να μην το έχει πετύχει ακόμα, αλλά αν μη τι άλλο είναι θέμα το οποίο συζητιέται ανοιχτά πια. Είναι θέμα σταθερότητας ενός συστήματος πολιτικού και κοινωνικού, το οποίο βέβαια είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κατάσταση μέσα στην οποία ζουν οι Κινέζοι στη χώρα τους. Μπορεί η συζήτηση πολλές φορές να είναι απογοτευτική όπως είπαν και ο κ. Μάν και η κυρία Μέσσα, αλλά παρόλα αυτά η συζήτηση αυτή πρέπει να συνεχίσει να γίνεται και να μην είμαστε αλαζόνες και να πούμε και αυτό και εκείνο και το άλλο. Όχι, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε εμείς και αυτό είναι η ελευθερία του συνδικαλίζεστε. Είναι πολύ σημαντικό γιατί εμείς αυτή η Επιτροπή είμαστε κοινωνικών υποθέσεων. Σε σχέση δηλαδή με τις διεθνείς δεσμεύσεις και τον διεθνή ρόλο της Κίνας, ε, σε αυτό πρέπει να κάνει κάτι. Πρέπει δηλαδή να τηρεί τις διεθνείς προδιαγραφές εφόσον είναι διεθνής παίκτη. Από εκεί και πέρα περιμένω τροπολογίες από τους συναδέρφους και θα δούμε. Ε, νομίζω ότι μπορούμε τώρα να περάσουμε στην ώρα της ψηφοφορίας. Εγώ τελείωσα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ λέει και η Προεδρεύουσα για την τελική σας τοποθέτηση για το θέμα αυτό και θα σας ευχαριστήσω εάν λάβετε υπόψη ότι όποιος θέλει να καταθέσει τροπολογίες θα πρέπει να το πράξει μέχρι τις 2 ε, Μαΐου στις, ε, το μεσημέρι. Και στη συνέχεια στις συνεδρίες 24-25 Μαΐου θα λάβουμε υπόψη αυτές τις τροπολογίες. Κλείνει αυτή η συζήτηση και περνάμε στις ψηφοφορίες. Η πρώτη έκθεση λοιπόν που πρέπει να τύχει ψηφοφορία είναι η έκθεση του κυρίου Ρίσσαρτ Φάουμπο για την εξωτερική διάσταση της ε, κοινωνικής πολιτικής. Νομίζω ότι έχετε τις ε, κάρτες ψηφοφορίες γιατί μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονικά μέσα. Όταν είναι απαραίτητο. Όταν είναι απαραίτητο θα το κάνουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με την τροπολογία 67 της κυρίας Τσίμερ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 69. Υπέρ, κατά, απόχες, απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 71 εκπίπτει εκπίπτει εγκριθεί σα στι 69 ναι, μπορούμε να την ψηφίσουμε παρόλα αυτά 71 ψήφι υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται 7 της ΔΕΒΕ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6, τροπολογία 73. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 74 και 75 είναι ταυτόσιμες. <clears throat> Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Παράγραφος 6 ε, ε, είναι τα δύο. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6α, τροπολογία 76, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7, τροπολογία 77, <clears throat> υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά, για να μην παραμείνει ίχνος αμφιβολίες. Αυτή την ψηφοφορία. Υπάρχουν δύο βουλευτέ που δεν έχουν κάρτα ψηφοφορία. Θα καταμετρήσουμε τις ψηφού τις, χειρο... τις τους χειρονακτικά. Κατά, 22 υπέρ, 19 κατά, εγκρίνεται τελικά. Η ε, 78. 78. Εκπίπτει. Τροπολογία 79. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 80 εκπίπτει στη συνέχεια. Παράγραφος 8. Ίντα 3. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9, η 81 απεσύρθη, παραμένουν οι τροπολογίες 82 και 83 που είναι και τα, τα φετώσιμες. Ψηφίζουμε. 82 και 83 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθησαν. 84 απεσύρθη. 85. Ψηφίζουμε. Όχι, όχι, γιατί ενεκρίθη 82. Οπότε εκπίπτει. Ψηφίζουμε την 85. Παρ' όλα αυτά ψηφίζουμε την 85. Ψήφι Κατά. Αποχές. Ας κάνουμε τον ηλεκτρονικό έλεγχο. Για την 85. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 85 πάντα. «32 με 10 εγκρίνεται» και μία απόχη «εγώ ήμουν αφηρημένη» λέει η πρόεδρος. 86, 87 και 88 είναι συμβατές με την 85. Θέτουμε σε ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Παράφος 10, τροπολογία 90, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97, υπέρ. κατά αποχές δεκτή. Είναι τα 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και φτάνουμε τώρα στην παράγραφο 11, συμβιβαστική τροπολογία Β, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, εκπίπτουν οι 92, 93, αλλά και 94. Περνάμε στην 106, στην παράγραφο 13, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική σε στην παράγραφο 12 ψήφι υπέρ <clears throat> κατά αποχές εγκρίνεται. Παρνάμε στην ε, συμβαστική δέλτα ψήφι υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Εκπίπτουν οι δύο επόμενες, πάμε στην 99 Ψήφι Κατά. Αποχές δεν γίνεται δεκτή. 98, 100 και 101 που είναι ταυτόσιμες. Ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Εκπίπτει 102. Πάμε στην 103 με χωριστή ψηφοφορία σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι κατά αποχές δεκτή δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 13 τροπολογία 105 και πάλι σε δύο τμήματα και 104 εξάλλου της εισηγήτριας του εισηγητή, συγγνώμη. Αλλά λόγω της έγκρισης προηγούμενης εκπίπτει και αυτή η τροπολογία. Πάμε κατευθείαν στην 107. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 108 εκπίπτει, 109 <clears throat> υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 110 εξέπεσε. Όχι, όχι, ψηφίζεται. 110. Ναι, ναι. Ψήφι υπέρ 110. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Θα ελέγξουμε. Για την 110. Για μένα ήταν σαφές το αποτέλεσμα. 110. Έλεγχος ηλεκτρονικό. Άρχεται η ψηφοφορία. Έντεκα υπέρ 33 ψήφοι κατά και με μία αποχή. Ήτανε σαφές. ΔΕΒΕ 4. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111 στην παράγραφο 15 ψήφι υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται. 112 στη διαπαράγραφο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Βεβαίως. Για την 112. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. 112 12 ηλεκτρονικός έλεγχος. Παρακαλώ. 38 υπέρ 7 κατά. Με τα τσαρούχια εγκρίνεται. Περνάμε. Οι 114 και 116 έχουν αποσυρθεί, παραμένει 115, στην παράγραφο 16 ψηφίσουμε την 115. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική F, σίγμα τάφ στα ελληνικά. Πάντα στην παράγραφο 16. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκπίπτουν οι 117 και 118, φτάνουμε στην παράγραφο 17, 119. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές υπάρχουν αφιβολίες οι οποίες πλανώνται και θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Αυτή την ψηφοφορία για την 119. «26 υπέρ, 20 κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται». Εκπίπτουν 120-121 Πάμε στη 17α, δβ 3 Ψήφι κατά, αποχές, εγκρίνεται. DV9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική ε, ε, ψήφι κατά, αποχές, εγκρίνεται εκπίπτουν οι άλλες δύο. Φτάνουμε στην ίντα 1, στην παράγραφο 17β, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 18, τροπολογία 123, ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Check. <clears throat> Έλεγχος 123, βεβαίως. 123 άρχεται η ψηφοφορία παράγραφος 18. «25 κατά και 22 υπέρ» απορρίφθηκε. Μεγάλο το δίκιο σας. 124. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα τρεις ταυτόσιμες τροπολογίες 125, 126, Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Πρώτη παράγραφος νέα, τροπολογία 68 σε δύο τμήματα. Συγγνώμη, το πρώτο τμήμα σε 68 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αλλά ας ελέγξουμε. Καλού κακού. Άρχεται η ψηφοφορία <clears throat> για την 68 τμήμα 1. 18 κατά, 29 υπέρ. κρίνεται Δεύτερο τμήμα της 68. Ψήφι υπέρ. Σήκωσε τα χέρια σας γιατί αλλιώς δεν μπορώ να βλέπω. Ψήφι κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Έγινε σαφές. Έλεγχος. Βεβαίως. Ό,τι θέλετε. 68 τμήμα 2. 68 δεύτερο τμήμα λοιπόν. «24 κατά και 23 υπέρ». Απερίφθη. Κάποιοι δεν ψήφισαν ή κάποιοι τροποποίησαν τη θέση τους. Ο ο Τόμας δεν έχει κάρτα και πρέπει να προσθέτουμε πάντα την δική του ψήφο στο, στο λογαριασμό. Απερίφθη, εν πάση Παράφος 18H είναι τα 10 ψήφι υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά έλεγχος ηλεκτρονικός για την 72 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται. 24 υπέρ, 23 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. 91 στην παράγραφο 10. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Είναι τα εννέα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 129. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φόη. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 129, παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίας. Ε, είναι μαλλον μάλλον. 35-9. Παράφος 15, τροπολογία 113, ψήφι πέρα. κατά αποχές εγκρίνεται. τα 4 ψηφιπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. τα 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 130 ψηφιπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Καλύτερα να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. 130. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκαεφτά, απορρίπτεται. 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά εγκρίνεται. Παράφορες 22, 136 απεσύρθη, 137, 138 και 139 που είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε λοιπόν την 137 με την 139 από κοινού ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 140 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΒ14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 143 προφορική με προφορική τροπολογία της κυρίας Μπερές σβήνει τα, τις λέξεις σε πλάγια στοιχεία, σε παχιά πλάγια, ψήφι περ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 23, τροπολογία 144, ψήφι περ κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Εκπίπτει 146 ή όχι. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, με συγχωρείτε. 146 υπέρ. Κατά. Ωραία, ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ίσως είναι καλύτερα. 146 ελέγχουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. E εγκρίθηκε 27 υπέρ, 19 κατά. 147 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 145 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Ε, παράγραφο 23, δεύτερο 12. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Παράγραφος 24, 149. 150 είναι παρόμοιες, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνονται. Και καταπίπτει 148, παράγραφος 24, 152. Υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές Απορρίφθηκε. Περνάμε τώρα στην παραγραφο 24153 υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίθηκε. Νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. 24154 υπέρ. Κατά απορρίφθηκε. Α, ε, αποχές απορρίφθηκε. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Προήμιο 4. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίθηκε. Τροπολογία 2 υπέρ κατά. Απόχες εγκρίθηκε. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αποσύρονται οι δύο επόμενες, 6 και 7. Περνάμε στην τροπολογία 8 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίθηκε. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Εντάξει, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να ελέγξουμε ηλεκτρονικά, μου λένε. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην 11. Τροπολογία 11. Η Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι 13 και 14 ε, αποσύρονται, 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17, 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται Απορρίφθηκε μάλλον, αλλά ας ελέγξουμε. Ψηφίζουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 17. Με ονομαστική κλίση. «18 υπέρ, 28 κατά». Απορρίφθηκε. Περνάμε τώρα στο συμβιβασμό, τροπολογία συμβιβασμού α. Υπέρ. Α, έκανα λάθος, με συγχωρείτε. Έχουμε την 18, με συγχωρείτε. 18 ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Τώρα περνάμε στην τροπολογία συμβιβασμού α. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν δύο επόμενες και περνάμε στην 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 25 και 26 είναι παρόμοιες και καταπίπτει 27. Περνάμε στην 30. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στις 28 και 29 καταπίπτουν 31, 31 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίφθηκε. 32, 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Τριάντα 33, 36, 34, 35, 38. Α, όχι, όχι. Ψηφίζουμε μόνο την 37. Οι άλλες καταπίπτουν. Μόνο την 37 ψηφίζουμε. Sim, Secretaria disse-me que iam as outras. Eh, estávamos só 37. 37 e e votos. Μόνο την 37 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην 39, η οποία ε, είναι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται της 39. Περνάμε στο J και τη 40, 41, 42 που είναι παρόμοιες. Υπέρ, κατά, απόχες, απορρίπτονται. 43 τρία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ. Α, με συγχωρείτε, είχα ε, ζητήσει να αποσυρθεί γιατί δέχτηκα το συμβάσμα. Πολύ ωραία, λέει η πρόεδρος, άρα αποσύρεται η 44 και φτάνουμε στο συμβιβασμό G. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και καταπίπτουν οι επόμενες, άρα περνάμε στη 48. Υπέρ, κατά, αποχές καλύτερα να επαληθεύσουμε, διότι υπάρχουν αμφιβολίες. Λοιπόν, 48 στην αιτιολογική σκέψη Κ, 48. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε με 26 ψήφους υπέρ και 19 κατά, 20 μάλλον, γιατί λείπει και μια κάρτα. Περνάμε στη 49. Υπέρ, κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά υπάρχουν ε, κάποιες αμφιβολίες. Γι' αυτό προτείνω να επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία επί της 49. Πέρας. Και έχουμε 28 κατά και 17 υπέρ. Πράγματι απορρίφθηκε. 50. Α, όχι, όχι, όχι. Εκπίπτει, καταπίπτει. Περνάμε λοιπόν στην 51. Στο L. Α, όχι, έχει αποσυρθεί. Περνάμε στην 52. Η 51 έχει αποσυρθεί. Περνάμε στην 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 54 υπέρ κατά επίσης απορρίφθηκε. 55 υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς ψήφισε το ΕΛΚ. Εγκρίθηκε, εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. Λέει η γραμματεία, εντάξει. Επειδή μερικοί δεν ψήφισαν, δεν ήμουν σίγουρη, αλλά εντάξει. M56 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 57 υπέρ, κατά,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 Πέρας και εγκρίνεται το σχέδιο γνώμης με 36 ψήφους υπέρ και 11 κατά. Να συγχαρούμε τον συνάδελφο για την έκθεση αυτή. Λοιπόν, περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία που αφορά τη γνωμοδότηση της κυρίας ε, Σάια για τη δημογραφική αλλαγή και τις συνέπειές της για τη μελλοντική πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια γνωμοδότηση, πρόκειται για μια γνωμοδότηση. Ωραία, έχετε τους καταλόγους στον κατάλογο μπροστά σας. Μπορούμε να αρχίσουμε λοιπόν. ο Παράγραφος πρώτη, Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά απόχες, απορρίπτεται. Τρία, Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία έξι, Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τέσσερα που ε, είναι σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Ωραία, αν θέλετε επαληθεύουμε το δεύτερο τμήμα της 4. Ε, Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. 25 κατά και 19 υπέρ. Άρα απορρίπτεται. Έχετε δίκιο. Απορρίφθηκε το δεύτερο τμήμα. Εδώ δεν ήταν απόλυτα σαφές. Τώρα ψηφίζουμε στην πρώτη παράγραφο την τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές, δεν είναι καθόλου σαφές. Καλύτερα να ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση, η οποία και αρχίσει. E λοιπόν, ψηφίζουμε την 5. Πέρας. 41 ψήφοι υπέρ, 2 κατά. Εγκρίνεται. Στην πρώτη παράγραφο 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8, τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Περάμε στη, στο συμβιβασμό α, στην δεύτερη παράγραφο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην δεύτερη παράγραφο, 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στο συμβασμό Β υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην ε, παράγραφο 3, 19. 19, τμήματική, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές και απορρίφθηκε νομίζω, αλλά καλύτερα να επαληθεύσουμε. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία και αρχίζει, για το δεύτερο τμήμα της 19. Δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Πέρας, 27 υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην 20. Παράγραφος 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 18 επίσης σε δύο τμήματα υπέρ του πρώτου τμήματος γιατί έχουμε τμηματική και εδώ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές επίσης εγκρίθηκε. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 25 στην παράγραφο 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίθηκε 24, 23 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 27 υπέρ. Όχι λέει η πρόεδρος. Καταπίπτει και περνάμε στην 28. 28 υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στην 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Περνάμε τώρα στην παράγραφο 4 Συμβιβασμός Γ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Καταπίπτουν οι επόμενες και περνάμε στην 34. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παίρναμε τώρα στο συμβιβασμό δέλτα, δέλτα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παίρναμε τώρα στην 37, διότι οι άλλες έχουν καταπέσει υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 38 υπέρ. 38, 38 είπα λέει ο πρόεδρος.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 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές. Α, με συγχωρείτε, παραπήγα γρήγορα. Λοιπόν, υπέρ, υπέρ και πάλι κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά γίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση για το σχέδιο γνωμοδότησης, η οποία και αρχίζει, η ψηφοφορία αρχίζει. Ένα μέλος από... Έχουμε έναν υπεράριθμο από τους σοσιαλιστές. Α, ήρθε και ο πρόεδρός μας, καλώς τον. Εντάξει. Πέρας της ψηφοφορίας... Τώρα έχουμε το σωστό αριθμό. Δεν έχουμε υπεράριθμους. 41 υπέρ 2 κατά και 3 αποχές. Άρα εγκρίνεται να συγχαρούμε την εισηγήτρια. Euh, Σας προτείνω να συνεχίσουμε την ψηφοφορία μας αγαπητοί συνάδελφοι. Και περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι η ψηφοφορία της έκθεσης της κυρίας Τζάνα Λάμπερτ. 1-2. Πρόκειται για τη διαχείριση ανακυκλωμένων καυσίμων και ενεργών αποβλήτων. Μαζί, πιέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 61 της κυρίας Στάνιλοκ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62 της κυρίας Στάνιλοκ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 και 63 μαζί που είναι οι ίδιες, υπέρ, κατά, αποχές, να επαληθεύσουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα τη ψηφοφορία, 26 υπέρ, λέει η πρόεδρο, 22 κατά, μία αποχή, εγκρίνεται. 64 έχει αποσυρθεί, 13 και 65 τώρα που είναι ίδιες, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 66, 67, 28 έχουν αποσυρθεί. 14 και 69 που είναι διαγραφή τις ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 70 της κυρίας Στάνρουκ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15, 71, 72, 16 και 73 3 δεν είναι αποδεκτές, οπότε φτάνουμε στο συμβασμό Α, στο άρθρο 4 σημείο 2. Υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το 4-2 έχουμε δύο ίδιες τροπολογίες, 18 και 76 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 77, Τόμας Χάντελ, με προφορική τροποποίηση του εισηγητή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το 2 δεσέ, λέει πρόεδρος, δύο ίδιες, 76 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 80 Στάνβερκ υπέρ, κατά αποχές θα επαληθεύσουμε. Νομίζω ότι απορρίπτεται, λέει η Πρόεδρος. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορίας. 21 υπέρ, 26 κατά. Απορρίπτεται. 21 και 79 είναι ίδιες. Ψηφίζουμε υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 81, 82 δεν είναι αποδεκτές. Όχι, είναι σαφές το αποτέλεσμα, λέει η πρόεδρος. Ωραία. Να επαληθεύσουμε τότε. Να επαληθεύσουμε. Παρακαλώ, πιο αργά σας παρακαλώ να πηγαίνετε και δεν καταλαβαίνω τίποτα έτσι όπως ψηφίζουμε, έτσι όπως λέτε τα νούμερα. Καλά, θα επαληθεύσουμε και έτσι θα μπορέσετε να έχετε χρόνο στη διάθεσή σας. 21 και 79 λοιπόν. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Κάποιος δεν ψήφισε. Α, τώρα είναι εντάξει. Πέρα τη φοφορίας. 26 υπέρ, 23 κατά. Εγκρίνεται τελικά. Ήρεμα, εντάξει. 83 στάνδριο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 84 του κυρίου Σόγκορ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 5, σημείο 1, ε22 της κυρίας Ζιν και 85 τόμα Χάντελ που είναι ίδιες. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 86 Steinrück έχει ζητηθεί κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, member stages shall ensure democratic control υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, το υπόλοιπο του κειμένου δηλαδή υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 6 σημείο 3, τροπολογία 23, Λάμπερτ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 6, 3β, 24 και 87 τροπολογίες της κυρίας Λάμπερτ και του κυρίου Χάντελ που είναι οι ίδιες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 25 Λάμπερτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 καταπίπτει, όπως και το 89. Ψηφίζουμε την τροπολογία 90, Handel, υπέρ, κατά, αποχές. Θα επαληθεύσουμε, αν και νομίζω ότι εγκρίνεται. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις υποφορία. 26 υπέρ, 22 κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται 90. Τροπολογία 91. Καταπίπτει. Ψηφίζουμε συνεπώς τώρα την τροπολογία 92 της κυρίας Στάνδρου. Κιπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 93 του κυρίου Τόμας Χάντελ έχει ζητηθεί κατά τμήματα ψηφοφορία από το ΕΛΚ. Αρχή του κειμένου. Τα κράτη-μέλη μέχρι verified manners. Υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά αποχές εγκρίνεται. Το υπόλοιπο κείμενο τώρα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 της συζυγήτρες είναι συμβατή, κατά τμήματα. Μα αφού πρόκειται για το ίδιο πράγμα, λέει πρόεδρος, πώς γίνεται να είναι συμβατή. Πρώτο τμήμα. Member States μέχρι verifiable manner. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το υπόλοιπο κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 7 σημείο 3. Τροπολογία 27 της εισηγήτρες και 94 του κυρίου Χάντελ που είναι ίδιες υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνονται. Άρθρο 7 σημείο 4. Τροπολογία 28 της εισηγήτριας και 95 του κυρίου Χάντελ με έτοιμα για προφορική τροποποίηση από την ίδια την εισηγήτρια. Αντιτίθεται κανείς την προφορική τροποποίηση. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν το σύνολο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 7 σημείο 5, τροπολογία 96 του κ. Χάντελ υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 7, νέο σημείο 5, 97, σόγκορ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 8 σημείο 2, τροπολογία 98 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, the safety case μέχρι risks for workers. Υπέρ, παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το υπόλοιπο κείμενο υπέρ, κατά. Οι φιλελεύθεροι τι κάνουν εκεί, δεν βλέπω, λέει πρόεδρος. Θα επαληθεύσουμε για το δεύτερο αυτό τμήμα. Α, σηκ, σηκώστε χέρια, ναι, υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 30, καταπίπτει. Και φτάνουμε στο άρθρο 8 σημείο 4, τροπολογίες 31 της εισηγήτριας και 99 του κ. Χάντελ που είναι οι ίδιες, ψηφίζουμε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Άρθρο 8, σημείο 4α, 2 ίδιες τροπολογίες, 32 και 100 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Άρθρο μετά το άρθρο 8 έχουμε τροπολογία 101 της κυρίας Στάνριουκ με προφορική τροποποίηση. Δεν είναι κανείς κατά ε, της προφορικής. Ωραία, άρα ψηφίζουμε την 101 τροποποιημένη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 102 της κυρίας Στάινμερ και πάλι προσφατοποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 9 συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έτσι φτάνουμε στο άρθρο 10, 108 τροπολογία του Χάντελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 39 λέει πρόεδρο καταπίπτει. 109 τώρα τροπολογία του άρθρου 11. άντελ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 12 σημείο 1. Συμβαστική γάμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 112 δεν αποδεκτεί. Άρθρο 14 τώρα, παράγραφος 1, σημείο 2. Ψηφίζουμε την τροπολογία 37 της εισηγήτριας με προφορική τροποποίηση. Δεν έχετε αντίρρηση για την προφορική τροποποίηση. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 14, παράγραφος 1, σημείο 7, τροπολογίες 38 και 114 που είναι ίδιες. Υπέρ, παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνονται. Ετυλογική σκέψη 1. Τροπολογία 42. Στάνριο και υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ετυλογική σκέψη 2. Τροπολογία 43. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ετυλογική σκέψη 3. Τροπολογία 44. Κυρία Στάνριο και υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την ετυλογική σκέψη 3. 46. Τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την λογική σκέψη 3. Ναι, να επαληθεύσουμε αν θέλετε. Επαληθεύουμε για τροπολογία 46. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 23 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογίες 2 και 45 που είναι οι ίδιες ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται μετά το ολική σκέψη 3 πάντα, 47 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 48 της κύριε Στάνουκ πάντα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την ολική σκέψη 19, τροπολογία 49 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ετρολογική σκέψη 27, τροπολογία 3 και 50 που είναι ίδιες, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνονται. Μετά την αλλογική σκέψη 27, τροπολογία 4 τη εισηγήτριας και 51 του κυρίου Χαντέλ, που είναι ίδιες υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Ευλογική σκέψη 29, Τροπολογίε 5 και 52 δεν είναι αποδεκτέ. Ψηφίζουμε τώρα στην αιτιολογική σκέψη 30 τις τροπολογίες 6 και 53 που είναι ίδιες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Μετά την λογική σκέψη 34 έχουμε την τροπολογία 7 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 Handel καταπίπτει. Ψηφίζουμε την 8 τώρα της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 κατά καταπίπτει. 56 του κύριου Χάντελ τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, μη λέτε έλεγχος αν δεν έχω πει ποιο είναι το αποτέλεσμα. Μετά την εντολική σκέψη 39 έχουμε την τροπολογία 9 της εισηγήτρες και 58 του κυρίου Χάντελ που είναι ίδιες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Εντολική σκέψη 41, τροπολογία 10 και 59 είναι ίδιες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Αιτιολογική γνώμη 1. Τροπολογίες 1 και 39. Του ζευγαριού Λάμπερτ Χάντελ που είναι ίδιες. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνονται, αλλά για να επαληθεύσουμε καλύτερα. Ηλεκτρονική ψηφοφορία 1 και 39. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της προφορίας. 25 υπέρ, 23 κατά εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Μετά την λογική γνώμη 1, τροπολογία 40 της κυρίας Στάνιρουκ. Καταπίπτει όμως αυτή. Οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία 41 της κυρίας Στάνιρουκ. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το σύνολο του κειμένου. Ηλεκτρονικά κύριε Σέρκας, Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 44 υπέρ, 4 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην ε, εισηγήτριά μας, την κύριε Λάμπερτ. Δεν είναι, αλλά ε, το θετικό πνεύμα θα φτάσει σε αυτήν. Και περνάμε στην τελευταία ψηφοφορία που έχουμε για σήμερα το πρωί και έχει που αφορά την προφορική ερώτηση και το ψήφισμα που προτείνουμε στην Ολομέλεια για την σύμβαση της ΔΟΕ για τους οικιακούς εργαζομένους. Όχι στα σπίτια όμως, αυτούς που δουλεύουν στα σπίτια. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί υπήρχε μια συζήτηση με τον κύριο Φάλμπρ για όλους αυτούς που καλύπτονται από αυτό το σχέδιο σύμβασης. Λοιπόν, θέτω σε ψηφοφορία. <clears throat> το, τη συμβαστική τροπολογία της εισηγήτριας όλο το κείμενο λοιπόν στη συμβαστική τροπολογία. Το σύνολο της προφορικής ερώτησης σε συνέπεια ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η προφορική ε, ερώτηση με τέσσερις ψήφους κατά. Τώρα, το κείμενο συμβιβαστικού χαρακτήρα για το ψήφισμα. Το σύνολο του κειμένου, όπως έχει τροποποιηθεί, χωρίς την αιτιολογική σκέψη Δέλτα, την παράγραφο 5, ούτε την παράγραφο 8. Ψήφι υπέρ. Με αυτές τις εξαιρέσεις. Ηλεκτρονικά. Ο Τσάμπα είναι υπέρ. Ο συντονιστής. Άρχεται. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 42. 43 υπέρ. 5 κατά καμία αποχή. Εγκρίνεται το κείμενο. Περνάμε τώρα στις τρεις επόμενες ψηφοφορίες. Χωρίς τα ψηφίζουμε. Αιτιολογική σκέψη δέλτα. Τις λέξεις on τις λέξεις προτείνεται να προσθέσουμε δύο φορές τη λέξη undocumented, άχαρτη, χωρίς έγγραφα δηλαδή. Μα αν δεν συμφωνείτε καταψηφίζετε και καταψηφίστε και ηλεκτρονικά κιόλας. Άρχεται η ψηφοφορία για την προσθήκη της λέξεως undocumented στην αιτιολογική σκέψη δεν. Άρχεται. Ποιο δεν ψήφισε. Ποιο δεν ψήφισε λέει η Ωραία, ψηφίσατε όλοι. 24 υπέρ, 23 κατά, εγκρίνεται η λέξη αυτή undocumented. Δύο φορές μάλιστα. Παράγραφος 5, προσθέτουμε τις λέξεις ελάχιστε αποδοχέ. Άρχεται η ψηφοφορία πάλι ηλεκτρονικά για την προσθήκη των λέξεων ελάχιστες αποδοχές, ελάχιστη μισθή. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. 18 υπέρ, 26 κατά, 2 αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 8. Ψηφίζουμε την τροποποιημένη μορφή του κειμένου με ηλεκτρονικό τρόπο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 19 υπέρ, 28 κατά. Δεν γίνεται δεκτή αυτή η παράγραφος 8 και ψηφίζω επομένως την τροπολογία 48 της κυρίας Άρκιν. Ψήφι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 48 Άρκιν γίνεται δεκτή με τρεις ψήφους κατά και θέτουμε τώρα το σύνολο του ψηφίσματος με ηλεκτρονικά μέσα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 40 υπέρ κατά, χωρίς αποχές. Ευχαριστούμε λοιπόν. Και θα υπάρξει επομένως συζήτηση στην Ολομέλεια για το θέμα αυτό στην επόμενη σύνοδό μας του, του, του, του Μαΐου, του Μαΐου λέει η Euh, Κλείσαμε τις ψηφοφορίες. Θα διακόψουμε τις εργασίες μας για να οργανωθούμε καλύτερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας προτείνω να σταματήσετε. Τι συνάδελφοι, σταματήστε τα πηγαδάκια, συγκεντρωθείτε. Έχουμε τελειώσει ψηφοφορίες. Et, Monsieur le Président, je... Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Συγγνώμη για την αταξία στην αίθουσα, αλλά νομίζω ότι τα έχετε συνηθίσει αυτά. Με τις κοινοβουλευτικές πρακτικές μετά από μια ψηφοφορία υπάρχει πάντα μεγάλη βαβούρα και δυσκολευόμαστε να οργανώσουμε και πάλι την κατάστασή μας. Αλλά η ποιότητα της ε, συζήτησης που οργανώνουμε δεν θα θυγεί από όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας. Γιατί είστε από την αρχή του χρόνου αυτού εκλεγμένος πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την κοινοβουλευτική μας Επιτροπή γιατί όταν, προβλέπουμε, όταν βλέπουμε τις επιτροπές οι οποίες προβλέπονται από τις συνθήκες υπάρχουν πολλές επιτροπές σε τεχνικό επίπεδο αλλά και αυτή για την κοινωνική προστασία και φυσικά λαμβάνει υπόψη η Εκτελεστική Επιτροπή την πολλαπλότητα ή την διτότητα τουλάχιστον των ερωτημάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ο προκάτοχός σας ερχόταν τακτικά στην Επιτροπή μας και έχει γίνει τώρα μια μικρή διακοπή παρουσίας, αλλά εγώ θα ήθελα να μπορέσουμε να επαναφέρουμε αυτή την τακτική πρακτική τουλάχιστον μια φορά το χρόνο <clears throat> να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων μαζί σας για να μας παρουσιάσετε την κατάσταση των εργασιών στα πλαίσια της τόσο σημαντικής αυτής της Επιτροπής που καθοδηγείται σε ένα τομέα πολύ σημαντικό. Έχετε το λόγο λοιπόν να μας, για να μας πείτε ποια είναι τα στοιχεία της επικαιρότητα στην Επιτροπή της οποίας προείσταστε και επίσης να μας εξηγήσετε πώς αξιολογείτε μέσα στην Επιτροπή αυτή την λειτουργία της ανοιχτή μεθόδου συνεργασίας καθώς και το γενικό πλαίσιο στο οποίο έχουμε ενταχθεί με τη στρατηγική 2020. Σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ απείρως κυρία Μπερές που μου δίνετε το λόγο. Θα μιλήσω πρώτα στα αγγλικά και αν έχετε ερωτήσεις θα απαντήσω στην δική μου την Ολλανδική μητρική γλώσσα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι εδώ παρόν και να παρουσιάσω την Επιτροπή κοινωνική προστασία τη Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχω την τιμή να προεδρεύω αυτή από την 1η Ιανουαρίου ενεστώτος. Πρέπει να πω καταρχήν ότι στα πλαίσια τη πληροφόρηση και τη διάδραση μεταξύ μα είναι πολύ σημαντική αυτή η ευκαιρία και θα χαρώ πολύ να επανέλθω και να σας ξαναδώ μια φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο όσο θέλετε και μπορούμε και εγγράφως φυσικά να σας διαβιβάσουμε πληροφορίες εφόσον το επιθυμείτε εσείς. Τα πρώτα μου σχόλια θα ήταν ότι πρέπει να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα και το εξάμεινο αυτό που επέρχεται για την Ευρώπη του 2020. Θα πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα την αξία των συστημάτων κοινωνική προστασία τη Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά διότι καλύπτουν με μία σπίδα τους πολίτες και τους εργαζομένους μέσα στην χρηματοοικονομική κρίση και έχουν δείξει μια μεγάλη ανθεκτικότητα παρά την διεθνή χρηματοοικονομική και οικονομική κρίση. Παρά, τα προβλήματα λοιπόν που αντιμετωπίζουμε στις οικονομίες μας σήμερα, τα κοινωνικά θέματα μέχρι στιγμής δεν έχουν ενταχθεί επαρκώς στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Η Επιτροπή μου πιστεύει ότι πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των χρηματοοικονομικών, οικονομικών και κοινωνικών πτυχών της στρατηγικής αυτής. Και παραθέτω εδώ. Θα επανέλθω στην συζήτηση. Μια σημαντική φράση σε ένα από τα κύρια μηνύματα που έχουμε στείλει εμεί στο Συμβούλιο και λέει τα εξής. Οι τροτότεροι θα πρέπει να προστατευθούν μέσα στα πλαίσια της εδραίωσης της ε, μεταρρύθμισης το, της κοινωνικής προστασίας ώστε να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα της κοινωνικής προστασίας και να συνδυάσουμε τις προσπάθειες των κρατών μελών μέσα στα πλαίσια αποτελεσματικότητας αλλά και αποδοτικότητας. Πρωτού έρθω στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής μας για να σας πω τι κάνουμε, να σας εξηγήσω την λειτουργία και τη φύση της Επιτροπής μας. Όπως φαίνεται η Επιτροπή Κοινωνική Προστασίας είναι ένα συμβουλευτικό σώμα που προβλέπεται από τις συνθήκε Άρθρο 160 για να παρακολουθήσει την κοινωνική κατάσταση και τι πολιτικέ κοινωνική προστασία, να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα αυτό και τι βέλτιστε πρακτικέ μεταξύ κρατών μελών και τη Κομισιόν. Η Επιτροπή Κοινωνική Προστασία δεν είναι πολιτικό σώμα. Πολιτικέ αποφάσει παίρνονται αλλού από το Συμβούλιο και από την Κομισιόν βασιζόμενοι όμως στην εμπειρία συσσωρευμένη εδώ και 10 χρόνια στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και των πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης, η Επιτροπή μας συμβάλλει για τα θέματα του Συμβουλίου Απασχόλησης και την κοινωνική διάσταση. Όπως λέει η συνθήκη, περιλαμβάνει εκπροσώπους των 7 27 κρατών μερών και της Κομισιόν Επιτροπή μας. Εμπλεκόμεθα σε όλες τις ε, πτυχές της κοινωνικής πολιτικής, υγειονομική περίθαλψη, κοινωνική προστασία και παροχές και αντιμετωπίζουμε και τις πολιτικές κοινωνικής συμπερίληψης, κοντολογής. Στέκομαι ή μάλλον κάθομαι σήμερα εδώ, όχι ως ένας πολιτικός ή δημόσιος υπάλληλος, αλλά ως κάποιος ο οποίος είναι προσιλωμένος στην επίτευξη περαιτέρω προόδου και συνεργασία στον τομέα αυτό για την ασφάλεια κτλ. των πολιτών σε κοινωνικό επίπεδο. Το Δεκέμβριο τον περασμένο εγκρίναμε το πρόγραμμα εργασίας μας και υπάρχουν ορισμένα θέματα που βρίσκονται στην ημερησία διάταξη που θα μας απασχολήσουν για εφέτος αλλά και του χρόνου. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η Επιτροπή μας θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τον κοινωνικό αντίκτυπο της οικονομικής και χρηματοοικονομικής κατάστασης και, την, και της συνεχιζόμενης παγιοποίηση των δημοσιονομικών των κρατών μελών και λαμβάνει υπόψη του μακροπρόθεσμου δείκτες και τι επιπτώσει για την κοινωνική προστασία και προκοπή. Αυτά θα περιλαφθούν και στην περιλαμβάνονται μάλλον συγγνώμη και στην πρώτη μας έκθεση για την, για την παγιοποίηση των κοινωνικών ζητημάτων μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020 που εκδόθηκε το Φεβρουάριο. Θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε επίση την επίτευξη των στόχων για την καταπολέμηση τη ένδυα και την κοινωνική συμπερίληψη, λαμβάνοντα πάντα υπόψη τις κατευθυντήρες γραμμές για την προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης και της καταπολέμησης της επάρατης ένδυας. Θέλουμε να συμβάλλουμε προς την ε, κατεύθυνση των συστάσεων για την αντιμετώπιση της ε, ένδειας από την Κομισιόν για τις συντάξεις. Η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας θα δώσει συνέχεια στις ε, αποφάσεις του Συμβουλίου για βαθύτερη μεθοδολογική ανατομή του τομέα αυτού και οι διαστάσεις αυτές του θέματος είναι φυσικά τμήμα των στρατηγικών που ενέκρινε το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα είμαστε σε επαφή επίσης με την Επιτροπή που ασχολείται για, με τις συντάξεις για την έκθεση γύρανσης του 2012. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η δυνατότητα των συντάξεων να συμβάλλουν στη μείωση της ένδυας. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική πτυχή του έργου μας. Οι συντάξεις δεν είναι μονάχα ένα σημαντικό θέμα σε οικονομικό επίπεδο λόγω της αύξησης του τμήματος του πληθυσμού που απολαμβάνει αυτόν, αλλά θα ήθελα να τονίσω το πιο σημαντικό γιατί οι συντάξει είναι ένα σημαντικό παράγον στο να εξαλειφθεί η ένδια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή μα στα πλαίσια τη έκθεση γύρανση ήταν κεφαλαιόδε, γιατί τόλμησε στο βαθμό δυνατού, δυνατού την κοινωνική διάσταση των συντάξεων. Στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και ξέρω ότι και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σας είναι ιδιαίτερα πρόσφυλες και συχνά στην μέση διαταξή σα, Θα συνεχίσουμε το έργο μας για την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ομάδα εργασία που θα αρχίσει να λειτουργεί σε μερικέ εβδομάδε. Η ομάδα εργασία θα εξετάσει τον, κύριο, νέο οδηγό για τι δημόσιε βοήθειε και τι δημόσιε προμήθειε που έχει προετοιμάσει η Επιτροπή μα πέρυσι. Θα αναλύσει επίση τις, ε, τα συμπεράσματα του τρίτου φόρουμ τη Επιτροπής Κοινωνικής Προστασία και θα συνεχίσει τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση των κρατικών κανόνων επιδότηση και η Επιτροπή μας θα παρουσιάσει τον Ιούνιο μία γνωμοδότηση για το πώς μπορούμε καλύτερα να παρουσιάσουμε τους στόχους μας στο νέο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Είπατε κυρία Πρόεδρε αν θα μπορούσα να πω κάτι για το θέμα αυτό. Αυτό μπορώ να σας πω ότι έχουμε προς στιγμή ε, μια ομάδα ad hoc με την προεδρία του Γάλλου συναδέλφου μας που εργάζεται σκληρά για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα μπορούμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες μας και ο στόχος μας είναι από τον, μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό του Ιουνίου να έχει περατωθεί αυτή η διαδικασία επί τη βάση και της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών. Θέλω να υπογραμμίσω περαιτέρω τη σημασία που επέχει η αμοιβαία μεταλαμπάδευση γνώσεων με, τις, ε, με τους ελέγχους ομοτήμων στα πλαίσια του Κομισιόν. Η Επιτροπή μας επίσης θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην πλατφόρμα κατά της ένδυας και του κοινωνικού ε, αποκλεισμού και έχουμε εγκρίνει ένα έγγραφο προβληματισμού για τη συνέχεια της ε, πολιτικής συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και εδώ ζητούμε να υπάρξει μια πλήρης ευθυγράμμιση κοινωνικής πολιτικής συνοχής και τη, της πολιτικής Ευρώπης 2020 που θα πρέπει να δώσει απαραίτητους πόρους για την, για την ε, αντιμετώπιση της ε, ένδυας και τη μείωση της ιδίας αυτής της ένδυας. Τώρα σε ό,τι αφορά τη στρατηγική 2020 και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Όπως είπα προηγουμένως, έχουμε κάνει μια έκθεση παρακολούθηση για την κοινωνική κατάσταση και την ανάπτυξη των πολιτικών κοινωνική πρακτική και προστασία που αντιμετωπίζουν την κοινωνική διάσταση τη Ευρώπη 20 και 20. Η έκθεση αυτή έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Απασχόληση και θα δημοσιευθεί ω ο νουπο. Αναλύει το πώ η κοινωνική πολιτική προστασία και οι κοινωνικέ προστασίε μπορούν να ευνοήσουν τι πολιτικέ αυτέ και να συμβάνουν στη συνολική επίτευξη αυτή τη στρατηγική. Ίσως μερικά από τα κύρια μήνυματα λοιπόν μπορώ να σας πω που προέρχονται από αυτή την έκθεση. Πρώτον, ένας στους κάθε πέντε Ευρωπαίους βρίσκεται στον κίνδυνο ένδυας και κοινωνικής, κοινωνικού αποκλεισμού και 40 εκατομμύρια άτομα βρίσκονται σε κατάσταση πραγματικής ένδυας. Το να μπορέσουμε να βγάλουμε λοιπόν αυτά τα άτομα από την ένδυα και την κοινωνική ε, κοινωνικό αποκλεισμό για 20 εκατομμύρια ατόμων μέχρι το 2020, αυτό απαιτεί φιλόδοξα μέτρα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μέσα στη συνολική μας στατική θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της ένδυας. Και στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο κατέληξε στα συμπεράσματά του υπογραμμίζων ότι το συνολικό αποτέλεσμα το οποίο προβλέπεται δεν θα επιτύχει τους στόχους και το ποσοστό απασχολησιμότητας 75% του 20 20. Δεν θα επιτύχουμε λοιπόν με τον τρόπο αυτό το στόχο του να ε, βγουν 20 εκατομμύρια άνθρωποι από την Ένδια. Τονίζει η εκθεσή μας ότι οι πιο ευάλωτοι θα πρέπει να προστατευτούν από την ένδια και τον αποκλεισμό. Δεν θα υπενθυμίσω λοιπόν αυτά τα οποία είπα προηγουμένως. Το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να μειώσουμε τα προβλήματα τα οποία προέρχονται από την αλλαγή καριέρας για να υπάρξει και επάρκεια των συστημάτων συνταξιοδότησης. Η έκθεση επίσης αναλύει την ανάγκη της ενεργού στρατηγικής συμπερίληψης και καλύτερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας και στις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες για να ξεπεραστεί ο κοινωνικός αποκλεισμό και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών παροχών και επίσης να αυξήσουμε τη δυνατότητα ενίσχυσης του αντικτύπου τη κοινωνικής πολιτικής σαν τμήμα μια γενικότερης στρατηγικής ελέγχου αντικτύπου. Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή μου ανησυχεί. Ανησυχεί για μερικέ εθνικέ αντιπροσωπείε γιατί η ετήσια έκθεση ανάπτυξης δεν αντανακλά πράγματι τη στρατηγική της Ευρώπης 2020. Μήπως θα υπάρξει κίνδυνος να συρρυκνωθεί η εμβέλεια της στρατηγικής της Ευρώπης 2020 και μπορούμε να συνεχίσουμε την σκέψη αυτή στην επικείμενη συζήτηση. Πρέπει λοιπόν από το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμεινο να εξασφαλίσουμε τη σωστή θέση για την κοινωνική διάσταση και το δεύτερο εξάμεινο θα θέσει τις βάσεις για το μελλοντικό έργο της Επιτροπής μας και την επιτυχή εφαρμογή μεταξύ άλλων της κατευθυντήριας γραμμής 10 κλείνων, κυρία Πρόεδρε. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της ένδυας που αναφέρεται στη στρατηγική 2020 δίνει μια μεγάλη συγκεντρικότητα στο έργο της Επιτροπής μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα. Κοινωνική προστασία και συμπερίληψη αναφέρονται πολλές φορές ως δύο ακρογωνιαίοι λύθη και αγκονάρια της διαδικασίας κοινωνικής ανάπτυξης της Ευρώπης. Η στρατηγική 2020 προτείνει μια σειρά από μέτρα τα οποία δημιουργούν την προσδοκία οριζόντιας αντιμετώπισης για όλη τη διάσταση της κοινωνικότητος. Αλλά στην πραγματικότητα, σαφής και διάφανη διαδικασία που αντιμετωπίζει την κοινωνική διάσταση δεν υπάρχει και θα πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα και συμπεράσματα τα οποία θα είναι πρόσφορα για την επόμενη άσκηση. Η, η Επιτροπή μας θα διαδραματίσει τον πλήρω στην εφαρμογή και την παρακολούθηση της στρατηγικής που εμπλέκει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο βάσει των αρμοδιοτήτων της η συμβολή όλων των άλλων θα είναι πάρα πολύ θετική και τον Οκτώβριο του 2011, αν θέλει ο Θεός, θα έχουμε μια συνάντηση μετά από την πρώτη συνάντηση για τη σύμβαση κατά της Ένδειας. Και είμαι σίγουρο ότι η Πολωνική Προεδρία θα βρει έναν τρόπο, κυρία Πρόεδρε, να σας αποδώσει τον ρόλο που αρμόζει στην Επιτροπή σας. Αυτό θα είναι μια, πραγματικά μια μεγάλη ευκαιρία να συνεχίσουμε το έργο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 2011, Οκτώβριο 2011 θα γίνει η συνάντηση αυτή. Ε, Παρακαλώ. Ο Ρώσα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε σε διάφορα σημεία στα οποία ήθελα να αναφερθώ και εγώ. Πρώτα απ' όλα, είπατε ότι η απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά την φορολογική παγίωση, όπως ονομάζεται, λέει ότι το θέμα της ε, προστασίας των πιο ευάλωτων είναι και το στοιχείο κλειδί. Και αυτό είναι που με ανησυχεί αυτή η διατύπωση, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκτός αυτής της κατηγορίας των περισσότερων ευάλωτων. Αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία, ένας στους πέντε, όπως το είπατε κι εσείς, κινδυνεύει να βρεθεί στην ένδια. Εδώ είναι τα 14 εκατομμύρια ή οι πιο ευάλωτοι. Είναι τα 14 εκατομμύρια που κινδυνεύουν να βρεθούν ε, στην Ένδια. Συμπεριλαμβάνονται όλοι αυτοί στην κατηγορία των περισσότερο ευάλωτων. Γιατί από αυτό εξαρτώνται και οι στόχοι που θα πρέπει να υιοθετήσουν τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την ένδια. Ένα άλλο σημείο που με απασχολεί και με απασχολεί και το Κοινοβούλιο που προετοιμάζει τη στρατηγική για το 2020 είναι κατευθυντήρια γραμμή για την Ένδια. Όπως είπατε και εσείς, συμπεριλαμβάνεται στην κατευθυντήρια γραμμή για την απασχόληση, ενώ η Ένδια είναι κάτι ευρύτερο, είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα από την ένδια στην οποία καταλήγουν τα άτομα που βρίσκονται στην ανεργία. Είτε επειδή είναι πολύ νέοι, είτε επειδή είναι πολύ μεγάλοι. Οπότε, μήπως τελικά η Επιτροπή σας αυτή την διάσταση θα έπρεπε επίσης να τη λάβει υπόψη, γιατί οι πιο ευάλωτοι, ο ένας στους πέντε που βρίσκονται σε κίνδυνο να βρεθούν στην Ένδια και το γεγονός ότι ο στόχος μας για την ε, Ένδια βρίσκεται στην κατευθυντήρια γραμμή για την ανεργία στα πλαίσια στρατηγικής 2020. Πώς πρέπει να τα δείτε όλα αυτά. Αναφερθήκατε επίσης και στις ε, κοινοφελείς υπηρεσίες και την κοινωνική τους διάσταση. Είμαι εισηγητής για την γνωμοδότηση αυτή, η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Ξέρετε ίσως ότι μία από τις προτάσεις που κάνω στην έκθεσή μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει μία πολυδιάστατη task force και να λάβουμε υπόψη μας το ρόλο που έχουν οι διάφορες γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής και να δούμε πώς θα συμπεριληφθούν οι κοινωνικοί εταίροι, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, που βοηθούν στον τομέα των κοινοφελών υπηρεσιών και της κοινωνικής τους διάστασης. Να δούμε τι έχουν, πώς μπορούν να συμπεριληφθούν όλοι αυτοί μαζί με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας αυτό το ρόλο ακριβώς πρέπει να έχει. Αυτό που είπατε εσείς σήμερα το πρωί μου επιβεβαιώνουν ότι τελικά ο ρόλος σας στην πραγματικότητα είναι καθαρά συμβουλευτικός και δεν είναι αυτός που θα ήθελα εγώ για μια ομάδα υψηλού επίπεδου που θα έπρεπε να είναι πιο δυναμικός και να πιέζει για αλλαγές στον τομέα των κοινωνικών ε, υπηρεσιών κοινή ωφελία. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζουμε τις διάφορες αποφάσεις που λαμβάνονται στα διάφορα επίπεδα, υπάρχει ο πολιτικός ρόλος, αλλά η Επιτροπή σας, όπως λέτε και εσείς, δεν είναι πολιτικό σώμα. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας για αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω στα Ολλανδικά, αν μου επιτρέπετε, λέει ο κύριος Μπέιτς. Για την πρώτη σας ερώτηση, που έχει να κάνει με τον ορισμό της ένδυας, της φτώχειας. Εδώ πρέπει να δούμε σε εθνικό επίπεδο τι ισχύει, γιατί οι χώρες μέλη αυτόνομα αποφασίζουν γι' αυτό. Για τη στραγική 2020 ξεκινήσαμε από τις εθνικές κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η σειρά είναι αυτή, κράτη-μέλη και μετά ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει το άρθρο 48 της συνθήκης και εκεί πρέπει να βασιζόμαστε. Πάντως πρέπει να ξεκινάμε ως σημείο κίνησης να έχουμε την πραγματικότητα. Καταλαβαίνω ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα δίλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πάντως η συνθήκη λέει αυτά που λέει. Η κοινωνική διάσταση πρέπει να προβάλλεται στην στρατηγική του 2020. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι βασιζόμαστε στο δίλημα αυτό και λέμε ότι στην Επιτροπή μας υπάρχουν διαφορετικές ε, απόψεις για το πώς πρέπει να λύσουμε το δίλημα αυτό. Ε, ζητάω κατανόηση μια που έχουμε ξεκινήσει μόλις. Και από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε ευρύτερα για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε για να λύσουμε το δίλημα αυτό. Έρχομαι τώρα στην ερώτησή σας όσον αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες ε, ε, της κοινοφελής. Στην ε, Επιτροπή μας είναι πολύ ψηλά στην ημερήσια διάταξη αυτή η προβληματική. Σίγουρα πρέπει να προετοιμαστούμε για να υποστηρίξουμε τις θέσεις μας μέσα στο Συμβούλιο. Πάντως υπάρχει μια άτυπη ομάδα εργασίας που ετοιμάσαμε στην τελευταία μας συνεδρία. Είναι δηλαδή κάτι πολύ πρόσφατο, άτυπη όπως σας είπα, ομάδα εργασίας, η οποία εξετάζει την νομική βάση. Γιατί πιστεύουμε ότι έχει μεγάλη σημασία να μαθαίνουμε ένας από τον άλλον και να διαπιστώνουμε έτσι ποιες τάσεις υπάρχουν όταν ε, θέτουμε σε εφαρμογή τις ε, κοινωνικές υπηρεσίες κοινή ωφελία. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με την προετοιμασία του επόμενου φόρου που κάνουμε αυτή την εποχή. Για να δούμε με ποιο τρόπο θα συνδέσουμε τις εργασίες αυτής της άτυπης ε, ομάδας εργασίας με την Επιτροπή μας. Θα συζητήσουμε λοιπόν και έτσι θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Για την παρατήρησή σας τώρα. Πολύ σωστά. Είπατε ότι ετοιμάζετε μια έκθεση. Τη γνωρίζω Και εδώ όμω πρέπει να γίνει ευρύτερη συζήτηση, κάτι το οποίο θα κάνουμε και θα φροντίσουμε να έρθουμε σε επαφή και μαζί σα πολύ σύντομα. Ε, Η κυρία Όμεν Ράιτερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μπέιτς που ήρθε εδώ. Όντως είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα σας και από πλευρά της Ολλανδίας. Εγώ από την Ολλανδία προέρχομαι και γι' αυτό το λέω αυτό. Τώρα γι' αυτό που είπατε. Εσείς και το έργο σας είναι η καλύτερη εγγύηση για να βγει ο κόσμος από την ε, ένδια. Όντως πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα ώστε οι άνθρωποι να βγουν από την ένδια να αποκτήσουν δουλειά. Και για να γίνει αυτό, πέρα από τα περί της στρατηγικής για το 2020 και πέρα από την κοινωνική διάσταση που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται εκεί, πέρα από αυτά, πρέπει να υπάρχει και ένα άλλο μέσο που είναι το κοινωνικό ταμείο ή το ταμείο για τις ε, επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Είναι και αυτά δύο μέσα, δύο εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας που μπορούν να βοηθήσουν τις κοινωνίες μας να βγουν από τη φτώχεια. Αναρωτιέμαι λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο τι δυνατότητες βλέπετε εσείς, εμείς, επικεντρωνόμενοι περισσότερο σε αυτό το θέμα, τι περισσότερο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δεύτερον, εμείς, και το λέτε και εσείς εξάλλου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να κάνουμε λίγα επειδή την κύρια αρμοδιότητα την έχουν τα κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι στην έκθεση για τις συντάξεις ήταν πάρα πολύ δύσκολο στο να καταλήξουμε ποιες είναι οι σωστές συντάξεις, αν πρέπει να μιλάμε για μια ελάχιστη σύνταξη, αν πρέπει να μιλάμε για επικουρικές συντάξεις κλπ. Δυστυχώς όμως διαπιστώνουμε ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινή ωφελία στις χώρες μέλη είναι εντελώ διαφορετικές μεταξύ τους από χώρα σε χώρα. Οπότε είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε συμπέρασμα. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να προχωρήσουμε, να συζητάμε μεταξύ μας για αυτό το θέμα ευρύτερα. Δεν είναι δυνατόν ένα κομμάτι της ε, κοινωνίας να έχει υψηλέ ε, συντάξεις, έσοδα και ανάλογα τμήμα τη κοινωνία να μην μπορεί να ζήσει από τις συντάξεις του. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μπέτ, ευχαριστώ. Το ότι έρχεστε από την Ολλανδία και εσεί. σίγουρα <clears throat> δεν θα πρέπει να παίζει κανένα ρόλο. Εγώ έτσι κι ακολουθώ τον ε, ε, κοινό παρονομαστή στην ε, Επιτροπή μας. Και μιλάω εκ μέρους της Επιτροπής, ως πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και όχι ως Ολλανδός. Συμφωνώ όμως μαζί σας ότι πρέπει ε, να βρούμε τον τρόπο, τον καλύτερο τρόπο για να βγάλουμε τον κόσμο από τη φτώχεια. Και σε αυτό μπορούν να βοηθήσουν οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινή ωφελία. Ναι, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στην Επιτροπή μας ε, να συνεργαζόμαστε και μαζί σας. Έτσι κι αλλιώς, τα θέματα της ε, κοινωνικής ένταξης είναι θέματα πάρα πολύ σημαντικά και πραγματικά η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Δεν είναι απλό και εύκολο να βρούμε μία λύση που να ταιριάζει σε όλους. Για τα άλλα μέσα στα οποία αναφερθήκατε, όντως υπάρχουν. Εμείς ασχολούμαστε κυρίως με τη στρατηγική 2020. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, έχουμε και γνωμοδότηση για το Ταμείο Συνοχής. Σίγουρα η δικιά μας επιτροπή θα έπρεπε να είναι πιο ισχυρή και να εμπλεχθεί περισσότερο όσον αφορά τη στρατηγική για το 2020. Συμφωνούμε με αυτό μαζί σας. Τώρα για το ποια είναι μια σωστή και αξιοπρεπή σύνταξη. Είναι βέβαια μια περίπλοκη προβληματική αυτή. Και υπάρχουν διαφορές στις ε, χώρες. Και γι' αυτό και η συζήτηση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και που θα κάνουμε στη συνέχεια για τους δείκτες θα είναι μια περίπλοκη συζήτηση. θα έρθει στην ημερήσια διάταξη πολύ σύντομα. Και σε συνεργασία και με την οικονομική πολιτική μάλιστα. Μπορώ να προσθέσω κάτι κυρία Πρόεδρε, λέει η κυρία Μενράτερ, Μια μικρή φράση μόνο. Κάνετε τις εκθέσεις σας, έχετε σε βουλευτικό ρόλο, οι γνωμοδοτήσεις σας έχετε την εντύπωση ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιάνουν τόπο. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ρωτάτε. Ναι. Νομίζω πως πρέπει να απαντήσω ναι. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όταν υπάρχουν ε, σημαντικά προβλήματα από την Επιτροπή Ασφάλειας συζητιόνται και φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι γνωμοδοτήσεις μας. Κύριε Κρίστενσεν, πρωτού δώσω στον κύριο Κρίστενσεν να σας πεθυμίσω ότι ο ρόλος της Επιτροπής έχει να κάνει περισσότερο με το Συμβούλιο και λιγότερο με την Κομισιόν. Κύριε Κρίστενσεν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας και είχα μονάχα ένα ερώτημα σε σχέση με την έκθεση στην οποία αναφερθήκατε και η οποία θα δημοσιευθεί και η οποία περιγράφει την κοινωνική κατάσταση στα κράτη-μέλη. Είπατε ότι εδώ πρόκειται για ένα κομβικό τομέα μέσα στη στρατηγική 2020. Συνδέεται όμως αυτό και σε ό,τι αφορά την κοινωνική κατάσταση σε σχέση με τον χώρο εργασίας για τους μετακινούμενους εργαζόμενους και αυτούς που μπορεί να περιγράψει κανείς ως οι εργαζόμενοι φτωχοί, οι οποίοι έχουν μεν μια θέση εργασίας, αλλά είναι τόσο χαμηλές οι αποδοχές τους, ώστε παραμένουν στα πλαίσια της ένδυας. Αντιμετωπίζει η και αυτά τα θέματα. Eh, Όσον αφορά την προβληματική αυτή της μετανάστευσης, νομίζω ότι δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα αυτή. Για την ένδια είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας. Το θέμα είναι να υπάρχουν οι σωστές διαδικασίες. Δεν μπορώ να σας πω σήμερα σε τι βαθμό ε, θα συμπεριλαμβάνεται η προβληματική αυτή στη δικιά μας γνωμοδότηση, αλλά θα συμπεριλαμβάνεται. Κύριε Ντερόσα, θέλετε και πάλι το λόγο. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ μία σύντομη παρατήρηση. Απαντών στην κυρία Όμεν Ρόιτεν, νομίζω ότι συμφωνήσατε ότι το θέμα της απασχόλησης ε, βρίσκεται μέσα στα πλαίσια της λύσης για την ένδια. Εγώ δεν διαφωνώ. Μιλάμε για αξιοπρεπή και καλή απασχόληση, αλλά οι στατιστικές στην Ιρλανδία δείχνουν ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι εργάζονται, αλλά βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο ένδυας. Πρέπει να αντιμετωπιστεί λοιπόν το πρόβλημα αυτό <clears throat> Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι συνταξιδοτημένοι, γυναίκες κυρίως που λόγω της αποσπασματικής εργασίας του παρελθόντος ζουν σε ένδια γιατί είναι ανεπαρκή στις συντάξεις τους. Αυτό που θέλω να τονίσω ότι ελπίζω ότι η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας δεν περιορίζει την ενατένιση της ένδυας μόνο κάτω από τον φακό των κατευθυντηριογραμμών για την απασχόληση. για το ένα στα πέντε άτομα που βρίσκεται σε κίνδυνο ένδυας έχετε στατιστικές που να καταδεικνύουν πόσοι από αυτούς βρίσκονται στο χώρο εργασίας, πόσοι είναι συνταξιούχοι, πόσοι από αυτούς είναι παιδιά ή επικεφαλής μονογονικών οικογενειών. Και επίσης για αυτά τα 14 εκατομμύρια τα οποία είναι σε βαθιά ένδια, πόσοι από αυτούς βρίσκονται ακόμα στο χώρο εργασία, γιατί αν θέλουμε πράγματι να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ένδυας θα πρέπει να δούμε πού ακριβώς βρίσκονται οι ενδέεις και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα άτομα με στοχευμένες πολιτικές. Ευχαριστώ πολύ. για την προβληματική αυτή της σύνδεσης ε, ένδυας ε, με την ε, ανεργία. Πρέπει να δούμε λίγο τι, λέει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Αυτή είναι πιο αρμόδιοι για τον ορισμό ναι, της αξιοπρεπούς εργασίας. Και αυτόν ο ορισμός πρέπει να ισχύει. Υπάρχουν στατιστικά δεδομένα, ήδη. Δεν τα ξέρω απ' έξω να σας τα πω, αλλά άμα θέλετε μπορώ να τα βρω και να σας τα παρουσιάσω. Θα ήθελα... Θα ήθελα να παρεύω για δύο θέματα. Για τους μακροοικονομικούς δείκτες καταρχήν, οι οποίοι είναι υποεκπώνηση στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης. Όπως ξέρετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περατώνει την διαβούλευση και καταλήγει στην οριστική του θέση για τα ζητήματα αυτά. Αλλά η Επιτροπή μας για τα κοινωνικά και την απασχόληση έχει δώσει γνωμοδοτήσεις ιδίω σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των μακροοικονομικών ε, ανισομεριών και των απαραίτητων δικτών για όλα αυτά, για το βαθμολόγιο στο μακροοικονομικό επίπεδο κτλ. και ανησυχεί για το γεγονός ότι ο μόνος μέσα σε εισαγωγικά κοινωνικός δείκτης ο οποίος θα ληφθεί υπόψη καταρχήν είναι ο δείκτης που αφορά το μοναδίο κόστος εργασίας. Ένα κριτήριο που ξέρουμε και μας λένε και πολύ ότι δεν είναι το αποφασιστικό κριτήριο για να αξιολογήσει κανείς την ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών. Και εμείς ανησυχούμε για αυτά τα οποία έχουν καθοριστεί στη ότι για αυτά που έχουμε καθορίσει στη στρατηγική 2020, εάν δεν μπορέσουν μέσα από το βαθμολόγιο να εξασφαλίσουν τη σωστή παρακολούθηση αυτών των θεμάτων, τότε θα μείνει με νεκρό γράμμα η στρατηγική 2020. Και δεν ξέρω αν εσείς συμμερίζεστε αυτή την άποψη στην Επιτροπή σας και ποια είναι η άποψή σας για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να να θα μπορούσατε να ενισχύσετε λίγο περισσότερο τη θέση σας και να περάσετε ένα μήνυμα που να δείχνει ότι χρειάζονται περισσότεροι και ευρύτεροι δείκτες. Γιατί υπάρχει ένας πολύ πολύπλοκος μηχανισμός που περιλαμβάνεται σε ένα από τα έγγραφα τα οποία μας δώσετε. Είναι φανερό ότι η Επιτροπή σας μεν έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο στα θέματα αυτά, αλλά το ερώτημά μου δε είναι πώς θα εξασφαλίσετε να, για να είναι το θέμα αυτό μια ενασχόληση της Επιτροπής σας σε μόνιμο επίπεδο ή το δεύτερο ερώτημά μου έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στη μελλοντική προγραμματική περίοδο είπατε ότι θα πρέπει να είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η στρατηγική Ευρώπης 2020 και εδώ φυσικά υπάρχει μια πλειοψηφία μέσα στην Επιτροπή μας που υποστηρίζει τη θέση σας. Υπάρχουν όμως τα εξής ερωτήματα που τίθενται. Πρώτα απ' όλα, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα ε, υπηρετήσει τους στόχους που του έχουν τεθεί και δεν θα χρησιμοποιηθεί ως στόχος κυρώσεων που έχουν αναφερθεί σε σχέση με την οικονομική διακυβέρνηση και το δεύτερο ερώτημα, στην συζήτηση για τις εξαρτήσεις, την επιλεξιμότητα. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτή η επιλεξιμότητα θα έχει θετικό πρόσημο. Θα είναι επιλεξιμότητα για την εφαρμογή της στρατηγικής, αλλά όχι όπως είπα προηγουμένως, ένα εργαλείο κυρώσεων και κολασμού στα πλαίσια της παρακολούθησης αυτής η οποία θα γίνει κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε οικονομική αδικία και αναποτελεσματικότητα. Για την πρώτη σας ερώτηση. Τώρα, μόλις μπαίνω στη διαδικασία και δεν έχουμε προχωρήσει περισσότερο. είναι η προβληματική η οποία συζητιέται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Διαφέρει βέβαια εκτίμηση ανάλογα με το με ποια αντιπροσωπεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει κανείς. Πρέπει βέβαια να φτάσουμε σε μια ε, διάφανη διαδικασία που να μπορούν όλοι να παρακολουθούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταλήξουμε έτσι στη στρατηγική για το 2020. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, αυτό είναι θέμα των ε, πολιτικών Είναι κάτι που επίσης θα συζητήσουμε την επόμενη περίοδο. Για το κοινωνικό ταμείο τώρα. μια στιγμή. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι στο κατάλογο των δικτών δεν θα πείτε εσείς ότι χρειαζόμαστε ένα δίκτυ για την καταπολέμηση της ένδυας, για την απασχόληση των νέων. Δεν θα τροφοδοτήσετε εσείς κάπως τη συζήτηση για να πείτε ποιοι πρέπει να είναι οι δείκτες, ώστε να υπάρχει η κοινωνική προστασία που θέλουμε. Ο κύριος Βέτς. Έχουμε αυτή τη στιγμή δείκτες, οι οποίοι έχουν καθοριστεί δεν αποκλείεται η συζήτηση να ξαναγίνει για τους δείκτες και θα το κάνουμε προετοιμάζοντας τη νέα διαδικασία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το προβλέψω. Έχει να κάνει με το σε ποια στιγμή της διαδικασίας θα βρισκόμαστε κάθε φορά. Eh, Όσον αφορά το κοινωνικό ταμείο, έχουμε γνωμοδότηση για τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή μας δεν παρεμβαίνει στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διατυπώνουμε όμως κάποια σημεία που θεωρούμε ότι μπορούν να βοηθήσουν όσον αφορά την αναλλαγικότητα. Ευχαριστώ για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων γιατί θα έχουμε και άλλες, ε, ε, άλλα φόρα ή και άλλα θέματα που θα μας απασχολήσουν όπως η ΔΕΚΟ. Θα ήθελα να σε επισύρω την προσοχή ε, για την έκβαση, την πορεία των συζητήσεων. Βλέπω ότι την προηγούμενη εβδομάδα το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ μπαίνει στον πυρήνα των δικτών που θα ληφθούν υπόψη ως ε, κύριοι μακροοικονομικοί δείκτες στα πλαίσια των νέων μέσων οικονομικής διακυβέρνησης. Και στο άτυπο αυτό Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ της προηγούμενης εβδομάδας έγινε λόγος για έναν κατάλογο δικτών. Εδώ βλέπω μόνο ένα ε, δείκτη σε σχέση με το εργατικό δυναμικό κάτι το οποίο δεν αρκεί κατά την άποψή μας για να λάβουμε υπόψη τις κοινωνικές ανισότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε γενικότερες μακροοικονομικές ανισότητες. Επιτρέψτε μου, αυτή την εποχή έχουμε δείκτη για το adequacy sustainability το θέμα είναι κατά πόσο έχει τις επιπτώσεις που θέλουμε και μπορώ να φανταστώ ότι η Επιτροπή για τους δείκτες ε, θα κάνει συζήτηση και θα το ξαναδεί. Πάντως υπάρχει σας ευχαριστώ για αυτή τη διευκρίνηση και γνωρίζουμε ότι η Βελγική Προεδρία συνεισέφερε ουσιαστικά για να φτάσουμε σε αυτούς τους δείκτες και σε αυτές τις γενικότερες ενδείξεις, αλλά θα πρέπει να μπουν στους σωστούς διάβλους για να μπορέσουν να είναι χρήσιμοι αυτοί οι δείκτες. Εκεί τους χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για, μια, για αυτή την ανταλλαγή απόψε και θα τα πούμε μελλοντικά και θα μιλήσουμε και για, το, για τον Οκτώβριο, για τα γεγονότα του Οκτωβρίου, για αυτά που προβλέπονται για τον Οκτώβριο, όπως μας προείπατε. Φτάνουμε στο τελευταίο θέμα του πρωινού μας. Πρόκειται για την παρουσίαση από την Επιτροπή του Πιλωτικού Σχεδίου που αφορά την βιομηχανική αναδιάρθρωση και τη συνέχεια που έχει δοθεί. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Λεμπρέ. Έχετε το λόγο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ λίγα λόγια πριν δώσω το λόγο στους ε, συναδέλφους του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που έθεσαν σε εφαρμογή αυτό το πρόγραμμα, αυτό το σχέδιο. Το θέμα της αναδιάρθρωσης σχετίζεται με μία ενεξελίξη οικονομία και δεν αφορά αποκλειστικά την κρίση ή συγκυριακά στοιχεία. Τα αίτια της αλλαγής είναι καθαρά διαρθρωτικής υφής και έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Είτε πρόκειται για τον τομέα των νέων τεχνολογιών, της παγκοσμιοποίησης, της δημογραφικής εξέλιξης, της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών, των νέων προϊόντων ή των νέων ετοιμάτων. Όταν μιλάμε για αναδιάρθρωση, θεωρούμε και λαμβάνουμε υπόψη τις αλλαγές ως προς το εργατικό δυναμικό. Και συνολικά αυτά τα φαινόμενα έχουν έναν αναπόφευκτο χαρακτήρα, θα μπορούσα να πω. Πρόκειται για μια διαρκή διαδικασία, μια μόνιμη βάση και πρόκειται για ένα μόνιμο πλαίσιο, μια μόνιμη πλαισίωση για την εξέλιξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ευημερίας των πολιτών. Υπάρχει ένας επιμερισμός ανά το χρόνο και ανά αναπεριφέρεια, αλλά οι αναδιαρθρώσεις αυτές είναι αφορούν μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε και αρνητικό αντίκτυπο για μία περιφέρεια, για μία ομάδα εργαζομένων και μεσοπρόθεσμες συνέπειες για αυτή την περιοχή, την περιφέρεια για τους εργαζόμενους. Άρα μας απασχολούν τα εξής. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι ενδιαφερόμενοι, οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι εργαζόμενοι επιχειρήσεις, οι περιφέρειες θα μπορούσαν κάπως να προτρέξουν και να διαχειριστούν αυτές τις αλλαγές για να μειώσουν το κοινωνικό ενεχόμενο κόστος λαμβάνονταν υπόψη την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να μοιραστούμε αυτές τις πρακτικές, να διαδώσουμε τις καλύτερες και να τις προωθήσουμε ανά την Ευρώπη. Για να προσπαθήσουμε, για να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις, το 2008 Ελάβαμε το πιλωτικό σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δώσουμε, να δώσουμε εκκίνηση στο σχέδιο αρένας. Δεν έχω εδώ τις διαφάνειες, διότι οι συνάδελφοι από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας έχουν αναπτύξει αυτά τα στοιχεία. Αυτά ήθελα να πω εν είδη εισαγωγής και ε, λέει η Πρόεδρος, κατανοώ ότι η θέση εφαρμογή αυτού του πιλωτικού σχεδίου οργανώθηκε από το ε, Γενικό Κέντρο Κατάρτισης του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Έχουμε την εκπρόσωπο ή τους εκπροσώπους εδώ αυτού του πιλωτικού σχεδίου και θα σας δώσω το λόγο. Ε, δεν ξέρω ποιος θα τον λάβει πρώτος, η πρώτη, η κυρία Ρίτζη και ο κύριος Τόμλινσον. Ο κύριος Τόμλινσον θα λάβει το λόγο πρώτος. Είμαστε από το Διεθνές Γραφείο Κατάρτισης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και διενεργήσαμε αυτές τις μελέτες στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπό το πρόγραμμα Αρένας ε, είχαμε ένα γενικό έγγραφο υποβάθρου για να δούμε τα διάφορα μέσα που έχουμε για να προτρέξουμε και να διαχειριστούμε την αναθιάρθρωση. Αυτό, τα, αυτό το εθνικό ιστορικό που έχουμε από όλα τα κράτη-μέλη που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας προετοιμάστηκε από 27 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και τα δεδομένα αυτά τα συζητήσαμε σε 27 τριμερή σεμινάρια και μετά επικαιροποιήθηκαν τα στοιχεία με βάση τα δεδομένα των σεμιναρίων. Έχουμε και μια συγκεφαλαίωση που προετοίμασαν τρεις ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες για να δώσουμε μία συγκεφαλαίωση των δεδομένων. Είναι μία ανεξάρτητη, πρόκειται για μία ανεξάρτητη μεθοδολογία, όμως υπάρχουν περιορισμοί ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν από χώρα σε χώρα. Και γι' αυτό ακριβώς έπρεπε να αποτιμηθούν από τους δικούς μας εμπειρογνώμονες. Βεβαίω, τα σεμινάρια, αφορούν τι απόψει όσων συμμετείχαν. Ήταν τριμερείς έπρεπε να δώσουμε αυτή τη συγκεφαλαίωση και αντιμετωπίσαμε αρκετές προκλήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Η έκθεση καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Απρίλιο του 2009 μέχρι τον Ιούνιο του 2010 και περιλαμβάνει 76 μέτρα για να προτρέξουμε στην αναθεώρηση 11 μέτρα για τη διαχείριση της αναδιάρθρωσης. Έχουμε 88 case studies και 800 συμμετέχοντες στη συζητήση του σεμιναρίου και είχαμε 54 ιδιωτικές εταιρείες που συμμετείχαν σε αυτές τις κατά περίπτωση μελέτες. Οι μελέτες διενεργήθηκαν μέσα στα πλαίσια της χρηματοπιστωτικής κρίσης που άρχισε το 2008 όπως γνωρίζουμε και μέσα στα πλαίσια περιπτώσεων αναδιάρθρωση είχαμε να κάνουμε με ε, αύξηση της ανεργίας από 7% το 2008 μέχρι 10% πέρσι. Έπρεπε λοιπόν να εφαρμόσουμε τα κυβερνητικά μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, αλλά η κατάσταση της αγοράς εργασίας ε, διαφέρει άρδιν από χώρα σε χώρα, καθώς και ο δείκτης ανεργίας και οι απολύσεις σε 22 κρατημέλη υπήρχαν πακέτα αντιμετώπισης της κρίσης κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις χώρες σε δύο-τρεις ομάδες. Υπάρχουν οι χώρες που επικεντρώνουν την προσοχή τους σε ε, υπηρεσίες αγοράς-εργασίας, η μέτρα καθώς και υποστήριξη της αγοράς-εργασίας. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη τα μέτρα που προβλέπονται για την αγορά εργασίας είναι πολύ περιορισμένα. Υπάρχουν ε, επίσης μέτρα υπηρεσιών και μέτρων, μεταξύ των οποίων Ιταλία, Δανία ε, και Σουηδία. Και υπάρχουν χώρες όπως η Γερμανία που υποστηρίζουν τα μέτρα υπέρ της αγοράς εργασίας. Και τώρα θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο για να σας μιλήσω για τα μέτρα που είναι διαθέσιμα για να προτρέξουμε στην την αναδιάρθρωση, στην αναδιάρθρωση της Ευρώπης των 27. Αυτό ε, δεν είναι μια καθολική, δεν αποτελεί μια καθολική έννοια. Έχει ένα διαφορετικό σημασιολογικό πεδίο ανάλογα με τη χώρα και Υπάρχουν πρωτοβουλίες βέλτιστων πρακτικών που τίθενται σε εφαρμογή για τη συνεχή εποπτεία των τάσεων της αγοράς εργασίας και μέτρα για την υποστήριξη της μετάβασης αυτής για την δημιουργία θέσεων και δεξιοτήτων καθώς και καινοτομιών. Σε σχέση με την πρώτη ε, ομάδα και τις προβλέψεις, οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση μπορούν να μας δώσουν πολλές πληροφορίες για τις τάσεις της αγοράς εργασίας. Επίσης, στη Φιλανδία έχουμε ένα δίκτυο προβλέψεων και προβλέψεις για την αγορά εργασίας για, στην Εστονία, στην Πορτογαλία από το Παρατηρητήριο Εργασιακών Εξελίξεων. Επίσης, σε περιφερειακό επίπεδο έχουμε πολλά παραδείγματα στην τσεχική δημοκρατία και το σχέδιο ε, καινοτόμων εξελίξεων στην αγορά εργασίας στη Φιλανδία. Τα τελικά μέτρα αφορούν το, μέτρο έγκαιρης, ε, το πρόγραμμα έγκαιρης ε, προειδοποίησης, όπου ξέρουμε ποιες είναι οι κινήσεις στην αγορά εργασίας, καθώς και σχέδια σε σχέση με απολύσεις που επιτρέπουν να προβλέψουμε μία προηγμένη στρατηγική και στην Αυστρία, Λιθουανία, Πολωνία και Ιρλανδία έχουμε πολύ ενδιαφέροντα σχέδια. Τώρα αυτό μας ενδιαφέρει να προλάβουμε, να προτρέξουμε και να υποστηρίξουμε και τη μεταβατική περίοδο έτσι ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να ε, προβλέψουμε και επενδύσεις και καινοτομίες. Όσον αφορά την υποστήριξη των καινοτομιών, Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εμπειρίες για την ε, προώθηση δεξιοτήτων στην Ολλανδία. Έχουμε και την περίπτωση των ε, τεχνολογικών πουλς στη Γαλλία και ορισμένες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των καινοτομιών στη, στον ΜΜΕ στην ε, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Σλοβακία μεταξύ άλλων χωρών. Επίσης, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για τις επενδύσεις όπως το σχέδιο Σάριο στη Σλοβακία. Η υποστήριξη της μετάβασης σημαίνει και πρωτοβουλίες καθώς και περιφερειακές έτσι ώστε να ανταποκριθούμε σε περιφέρειες όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην αγορά εργασίας, υπάρχουν συγκεκριμένες εμπειρίες στον ε, τομέα της Ολλανδίας, στον κατασκευαστικό τομέα και στο, σε περιφερειακό ε, επίπεδο. Υπάρχει συνεργασία και συμμετοχή για να προωθήσουμε τις επιχειρήσεις αναπεριφέρειες όπως στην Ιταλία και την περιοχή Γκέτεμπορκ στη Σουηδία. Εκεί προβλέπεται ένα άλλο σχέδιο. Υπάρχουν, υπάρχει περιορισμένος αντίκτυπος βεβαίως που αφορά τις περιφέρειες. Η τελευταία ομάδα υποστήριξης των μεταβατικών δράσεων αφορά τους πολίτες γιατί οι αλλαγές ε, είναι πολύ πιο δύσκολες ε, για τους ε, ε, πολίτες, ιδιαίτερα για αυτούς που ήταν ε, εργοδότες ή εργαζόμενοι και ιδιαίτερα εργοδότες επί σειρά ετών. Μιλάμε για νέες ευκαιρίες και ηλικιακές ομάδες στην Πορτογαλία και το σχέδιο λογιστικών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η επαγγελματική κατάρτιση είναι πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες που δημιουργούνται με βάση τις απολύσεις. Στη Γερμανία έχουμε την διαβίου μάθηση των εργαζομένων, ένα ειδικό πρόγραμμα δηλαδή, και αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν να προωθηθούν, όπως στη Γαλλία στην περίπτωση συλλογικών συμβάσεων, μέσα τα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας στον χώρο εργασίας. Ποια είναι τα βασικά διδάγματα για την αντιμετώπιση, την έγκαιρη αντιμετώπιση. Είπαμε ότι δεν πρόκειται για μια καθολική έννοια, αλλά υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες και μέτρα τα οποία προβλέπονται. Μιλάμε για συλλογή δεδομένων και παρεπόμενες δραστηριότητες. Αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες για την εφαρμογή αυτών των μέτρων στα ΜΜΕ και αυτό που έχει σημασία είναι να προωθήσουμε συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης και σε ε, επίπεδο επιχειρήσεων μιλάμε για, για, το, για τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικές συμβάσεις, διαπραγμάτευση συλλογικών συμβάσεων. Τώρα, μιλώντας ε, για την ε, διαρθρωτική προσέγγιση. Μιλάμε για ε, μέτρα πρόληψης, δηλαδή να γι, μην γίνονται απολύσεις ή να καταπραίνουμε κάπως αυτά τα μέτρα ε, με τη μετάβαση σε νέες θέσεις εργασίας. Αυτά τα μέτρα έχουν εφαρμοστεί μαζικά κατά τη διάρκεια της κρίσης ως προς την πρώτη ομάδα μέτρων οι απολύσεις είναι ε, τελευταίο μέτρο στο οποίο καταφεύγουμε και υπάρχουν κοινά μέτρα που προβλέπονται, δηλαδή μείωση μισθών, επιδοτήσεις, μερική απασχόληση ή ε, προσωρινές απολύσεις. Ε, η μείωση των μισθών εφαρμόζεται σε πολλές χώρες, ε, αυτό αφορά και τα επιδόματα ή δεν υπάρχουν πια αποσπασμένοι εργαζόμενοι. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε μία συμφωνία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Θα πρέπει να δούμε ποιες επιδοτήσεις έχουν ε, πια επίδραση. Υπάρχει ένας μακρύς ε, κατάλογος κριτηρίων επιλεξιμότητας και πολλές φορές γνωρίζουμε ότι οι επιδοτήσεις χορηγούνται σε σε μη παραγωγικές ε, επιχειρήσεις που δεν έχουν προοπτικές για το μέλλον. Πολλές επιχειρήσεις έχουν ένα ευέλικτο χρόνο εργασίας, ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση Υπάρχει και περισσότερη εργασία. Μας ενδιαφέρουν ε, τα σχέδια της ε, Γαλλίας, Αυστρίας, Ιταλίας και Λουξεμβούρου επί του θέματος επιμερισμού εργασίας. Σε ορισμένες χώρες αυτές οι διευθετήσεις αφορούν κρατικές επιδοτήσεις για την αποζημίωση εργαζομένων ή αντισταθμιστικά μέτρα. Ένα από τα δύναμα σημεία είναι ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε την οικονομική ανάκαμψη με βάση τα σχέδια αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μερική απασχόληση, η μερική ανεργία. Μειώνουμε το χρόνο εργασίας με κρατικές επιδοτήσεις πολλές φορές, αλλά αυτά τα μέτρα μερικής απασχόλησης απολύσεις αφορά ε, μειώσει στο χρόνο εργασίας, αλλά σε πολλές χώρες θεωρείται μία αδύναμη προσαρμογή στην αυξανόμενη παραγωγή και σημαίνει ότι αναβάλλονται οι απολύσεις και τίποτα άλλο. Για να αποφύγουμε απολύσεις στο σύνολό προβλέπουμε προσωρινές απολύσεις. Έχει επίσης ε, μεγάλη σημασία το χρονικό πλαίσιο από χώρα σε χώρα. Μιλάμε για συγκεκριμένες ε, ομάδες εργαζομένων και τομέων. Πολλές πρωτοβουλίες έχουν ε, αναλυφθεί από το Βέλιο και την Ιταλία για ένα ταμείο εγγυήσεων και όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικές ως προς τις απολύσεις. Τα εξή μέτρα προβλέπονται πρόορη συνταξιοδότηση καθώς και μετάβαση σε εναλλακτικέ θέσεις εργασίας. Η πρώιμη συνταξιοδότηση είναι ένα κοινό μέτρο σε πολλά κράτη-μέλη και σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στην Ισπανία θεωρείται θεωρείται πλεονεκτικό μέτρο σε σχέση με ένα άνοιγμα ως προς ε, ενδεχόμενες νέες θέσεις εργασίας, αλλά είναι αμφιλεγόμενο σε σχέση με τη βιωσιμότητα των, ε, του συνταξιοδοτικού. Σε αρκετές χώρες έχουμε συλλογικές απολύσεις, αλλά αυτό ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα. Δεν υπάρχει όμως νομική υποχρέωση σε όλες τις χώρες, δηλαδή στη Δανία και τη Σουηδία και πολύ συχνά θεωρείται επιπρόσθετος φόρτος για τους εργοδότες για μια χρονική περίοδο. Το τελικό μέτρο, το Job Counseling, είναι το καλύτερο μέτρο μετάβασης μέσα στα πλαίσια των απολύσεων. Γίνεται από δημόσιους φορείς στη Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία. Υπάρχει μία, ένας αναδιόμενος ε, τομέας ε, που προβλέπει αυτές τις υπηρεσίες και στο Βέλγιο και τη Γαλλία υπάρχουν κοινωνικά συνοδευτικά σχέδια για να καταπραίνουμε τον αρνητικό αντίκτυπο των ε, απολύσεων. για να υποστηρίξουμε τη μετάβαση και την επανεισδοχή στην αγορά εργασίας. Αυτή η υποστήριξη έχει μεγάλη σημασία μέσω πρωτοβουλειών για να προωθήσουμε αρμοδιότητες, προσόντα μάλλον και δεξιότητες. βεβαίως η κατάσταση δεν είναι ίδια, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Υπάρχει η πιστοποίηση της εργασίας στην Εστονία σε σχέση με τη συνεχή κατάρτιση στην Ολλανδία, στην Τσεχική Δημοκρατία υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα και στην Πορτογαλία υπάρχει το πρόγραμμα επαγγελματικών προσόντων. Τέλος, τα βασικά διδάγματα αφορούν μια, ε, ένα ευρύ φάσμα μέτρων, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι πώς εφαρμόζεται ανα κράτος μέλος και μας ενδιαφέρει και η συμμετοχή του κράτους η οποία δεν είναι η ίδια. Πολλές φορές υπάρχει εκτενής ρύθμιση, κρατική ρύθμιση και τα μέτρα πολλές φορές είναι περιορισμένα σε σχέση με την κατάσταση της αγοράς εργασίας, ενώ σε άλλες χώρες τα ε, μέτρα, τα κρατικά μέτρα αφορούν κάθε μορφή αναδιάρθρωσης. Τα περισσότερα κράτη-μέλη θέλουν να αποφύγουν τις πωλήσει πρόθεσμα και μόνο ορισμένα κράτη δίνουν προτεραιότητα στην επαγγελματική μετάβαση για να εξευρεθούν ε, νέες θέσεις εργασίας παρά να υπάρξουν περικοπές στην, ε, στο μισθολόγιο. Επίσης, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς θα επεκταθούν αυτά τα ε, μέτρα κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά είναι δύσκολο να αποτιμηθεί ο αντίκτυπος. Έτσι η μελέτη αυτή καταδεικνύει την δυναμική και τις τάσεις οι οποίες διαγράφονται και όλα αυτά δείχνουν ότι ο κοινωνικός διάλογος είναι πάρα πολύ σημαντικός για να προκαταλάβει κανείς και να προβλέψει τις αναδιαρθρώσεις εφόσον φυσικά βασίζεται σε μια παράδοση αμοιβαία εμπιστοσύνη και όταν υπάρχει καλή επικοινωνία και καλό θεσμικό πλαίσιο. Οι κατοικές, ε, κρατικές παρεμβάσεις για τη διαφύλαξη των θέσεων σε οικονομικές κρίσεις ήταν σαφείς και ορατές σε πολλές χώρες και πολλά συστήματα τα οποία υπήρχαν επεκτάθησαν ή παρατάθηκαν. Υπάρχουν στοιχεία επίση καινοτομία στην υποστήριξη που δίδουν οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. Με στόχο να προλάβουν τις αλλαγές και να δράσουν εγκαίρως με ταχεία απάντηση. Υπήρξε περισσότερη εμπλοκή των αποκεντρωμένων κυβερνητικών δομών, τοπικής και αυτοδίκησης κτλ. για την ε, σχεδίαση της ε, οικονομικής μετα... μεταλλαγής και της ε, αναδιάθρωσης. Τα διλήμματα τα οποία προκύπτουν από τη μελέτη και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά είναι καταρχήν το θέμα της επιλεξιμότητας των ατυπικών και ε, προσωρινά εργαζόμενων εργαζομένων για υποστήριξη, η επιλεξιμότητα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες δημόσιας παροχής εργασίας, σε βάση μερικής απασχόλησης μονάχα, τις σχέσεις με κοινωνική προστασία και δικαιώματα σύνταξης. Επίσης, οι πρακτικές αναδιάθρωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις τείνουν να είναι πιο περιοριστικού χαρακτήρα από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και βασίζονται σε ουσιαστικά επιδόματα ανεργίας και αντιστάθμισμα για την απώλεια εργασίας και όχι επανακατάρτιση. Υπάρχουν ομάδες πληθυσμού που είναι τρωτές όπως είναι οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία Αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι συνήθως χάνουν κατά τη διάρκεια περίοδων αναδιάρθρωσης. Ένα από τα κύρια θέματα που εξετάστηκε είναι πώς να οριοθετήσουμε την ευθύνη της επιχείρησης εναντί του κράτους κατά τη διάρκεια της μετάβασης. Ποιος πρέπει να πληρώσει, ποιος έχει την ευθύνη. Το θέμα λοιπόν της επαναεκπαίδευσης ήταν πάρα πολύ σημαντικό σε όλα τα εθνικά σεμινάρια. Πολύ συζήτηση είναι για την αποτελεσματικότητα <clears throat> της ε, επαγγελματικής ε, εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης στην επιχείρηση για την παροχή δεξιοτήτων που ήταν απαραίτητες για να βρεθεί κανεί, κανείς πάλι με μια θέση εργασίας. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν στην ε, ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης για την ε, απασχόληση και επίσης του δικού μας φορέα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Σας ευχαριστούμε πολύ ο κ. Χρίστιανσεν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για τις παρατηρήσεις τους. Αναμφιβόλως ο τομέας αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη και να υπάρξει ανάκαμψη. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν την απαραίτητη αναδιάρθρωση και να ατενίσουν το μέλλον. Έχουμε πράγματι καλές ευκαιρίες, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι μικρές. Και έτσι μπορούν εύκολα να αναδιαρθρωθούν, να τροποποιήσουν τις παραγωγικές τους διαδικασίες και να τις προσαρμόσουν στην ζήτηση η οποία αναδύεται στην αγορά. Εγώ υπήρξα εισηγητής για την Εύελιξ Ασφάλεια το 2007. Τότε κάναμε κάποιες ε, συνεδριάσεις, μάλλον αποφασίστηκε σε κάποιες συνεδριάσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ότι η ευελίξη ασφάλεια με τη μία ή την άλλη μορφή θα πρέπει να εισαχθεί σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντα σε, ένα, ε, σε μία μορφή που ε, προσάδει στις ε, κοινωνικές συνθήκες και παραδόσεις των χώρων ε, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ορισμένες μαζί με τις συλλογικέ συμβάσεις. Στην Δανία ήταν ένα παράδειγμα αυτό. Άλλες χώρες χρησιμοποίησαν την νομοθετική μέθοδο για την προστασία των εργαζομένων. Εύελιξη ασφάλεια σημαίνει ευελιξία αλλά και κοινωνική ασφάλιση. Και εδώ Νομίζω ότι λείπει ακόμα κάτι στον τομέα αυτό. Γιατί δεν μιλάμε για την ε, μαζική και ενεργή επένδυση στις πολιτικές του χώρου εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Στη Δανία πάνω από 6% του ΑΕΠ μας δαπανάται για την ύπαρξη μιας ενεργούς πολιτικής στον εργασιακό χώρο. Αυτό το κάνουμε για να έχουμε και ευελιξία στην αγορά εργασίας, αλλά και ασφάλεια και έχουμε πολύ υψηλό επίπεδο κάλυψης όταν τα άτομα χάνουν τη θέση εργασίας, έρχονται για αρρωγή σε εμά, παίρνουν επιδόματα και όλοι οι άνεργοι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα ενεργό σχέδιο για το μέλλον τους, ένα σχέδιο υποστήριξης. Αν το κάναν αυτό όλες οι χώρες, δεν θα βρισκόμασταν στη σημερινή κατάσταση. γιατί εάν υπάρχει μεγαλύτερη ευκαμψία μπορεί ο εργαζόμενος να βρει πιο εύκολα θέση εργασίας. Δεν μπορεί να υπάρχει μόνο η ευκαμψία γιατί ο εργαζόμενος τότε δεν νιώθει καμία ασφάλεια. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα μιας εξασφάλισης ότι μετά από μια μεταβατική φάση αναπροσαρμογής θα μπορέσει τελικά ο εργαζόμενος να ξαναβρει δουλειά. Αυτό δεν γίνεται βέβαια όμως άμα δεν το θέλουν οι εργαζόμενοι ή τα συνδικάτα. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να χάσει κανεί τη θέση εργασία του. Ένα από τα θέματα που αναφέρατε στι ενισχυμένε δυνατότητε για συμβάσει περιορισμένου χρόνου στην αγορά εργασίας ή για μερική απασχόληση εργασίας ή για διαμερασμό θέσεων εργασίας ή για ε, εθελοντική μείωση μισθών. Εδώ μου λείπει κάτι στον τομέα της ε, συμμετοχής του εργαζομένου και θα προκύψουν πάρα πολλές συγκρούσεις εάν αυτή είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε και δεν υπάρχει πραγματική επένδυση στις δυνάμεις εργασίας για να υπάρξει η απαραίτητη ευελιξία και να γίνουν οι μεταλλαγές αυτές που χρειάζονται στο μέλλον για την ανταγωνιστικότητα με ομαλό τρόπο. Σας ευχαριστώ. αυτή την βόρεια άποψη. Τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι αφού προηγουμένως κάνω ένα σχόλιο μετά από αυτά που ακούσαμε από τον συνάδελφο. Γιατί, γιατί εγώ εκτιμάω όλος ιδιαίτερο το βόρειο σύστημα. Και καλό θα ήταν το ευρωπαϊκό σύστημα να εμπνευστεί από αυτό. Τότε θα μπορούσαμε να μιλάμε για ευελιξία και ασφάλεια κάτω από καλές συνθήκε. Αναρωτιέμαι όμως στην ουσία μήπως είναι αλήθεια ή όχι ότι μπορεί να μεταφερθεί τόσο εύκολα ε, στην Ευρώπη λαμβάνοντας υπόψη τη συνοχή. Θα ήταν ενδιαφέρον δηλαδή εσείς να μας πείτε κατά πόσο στην μελέτη σας βλέπετε να υπάρχει αυτή η διαφορά. Όσον αφορά την αξιολόγηση της αναδιάρθρωσης ανάλογα με την συνοχή ε, την κοινωνική που υπάρχει στη μία και στην άλλη περίπτωση. Θα επανέλθετε φαντάζομαι στην απάντησή σας. Ε, και μια άλλη παρατήρηση που έχω να κάνω. Ως Ευρωπαίος νομοθέτης, εμείς προχωράμε εξετάζοντας την υπόθεση βήμα-βήμα. δικιά μας ευθύνη όταν εξετάζουμε θέματα παρέμβασης του Ταμείου ε, που βοηθάει στις συνέπειες από την παγκοσμιοποίηση, ε, φροντίζουμε να κινητοποιηθεί σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης που βρίσκονται στα χέρια πολυεθνικών μερικές φορές. Εγώ θα έλεγα όμως ότι αντί να κινητοποιήσουμε το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, καλύτερα θα ήταν να έχουμε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία που να δεσμεύει τις πολυεθνικές να πηγαίνουν πιο μακριά από αυτά που περιλαμβάνονται στις συλλογικέ συμβάσεις και στις εθνικές νομοθεσίες. Εσείς λοιπόν, μετά από αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, μετά από αυτή τη μελέτη που κάνατε, καταλήγετε σε συμπεράσματα για πρωτοβουλίες που θα έπρεπε να αναλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο ξέρω ότι το πρώτο που θα μας προτείνετε είναι έναν κώδικα διοντολογίας. Εντάξει, αλλά μπορούμε να πάμε και πιο πέρα. Μπορούμε να επιμείνουμε στον Επίτροπο ώστε να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ή πιστεύετε ότι ζητώντα την κινητοποίηση των κοινωνικών εταίρων θα υπάρχει αυτός ο κώδικας. Ποια είναι τα αποτελέσματα δηλαδή μετά από αυτήν την ε, πιλωτική έρευνα, το πιλωτικό πρόγραμμα. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε, για την τελευταία σας ερώτηση μπορώ να σας ε, παρουσιάσω κάποια συμπεράσματα, κάποια πρώτα συμπεράσματα στο οποία καταλήξαμε μετά από την προσπάθεια αυτή που κάναμε εξετάζοντας την κατάσταση στις 27 χώρες. Είδαμε ότι υπάρχουν πολλές πρακτικές και καινοτόμες συχνά. Έτσι, η εικόνα είναι κάπως πιο ξεκάθαρη για το ότι μέσα διαθέτουν 27 χώρες μέλη. Η έκθεση που πήρετε συμπληρώνεται και από 27 τέτοιες εκθέσεις που αφορούν η κάθε μία από μία ευρωπαϊκή χώρα. Δεν υπάρχει λοιπόν ενιαία λύση, το είπαν και συνάδελφοι, υπάρχουν διαφορές. Όμως, αυτό που βγαίνει από την ανάλυση μας είναι ότι τελικά υπάρχει μια σύγκληση και υπάρχει μια κοινή προσέγγιση. Τουλάχιστον μια τάση προς μια κοινή προσέγγιση που λέει ότι χρειάζεται η επαγγελματική προσαρμογή. Αλλά με τεράστιες διαφορές ακόμα, εννοείται. Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αντιδραστικές αντιμετωπίσεις. Θα κλείσουμε, δεν έχουμε προετοιμαστεί, δεν γίνεται. Γι' αυτό και θέλουμε και την νομοθεσία που να προστατεύει από τις μαζικές απολύσεις. Εξακολουθούν όμως τέτοια φαινόμενα να είναι τραυματικά για πολλές περιφέρειες. Τώρα ρωτάτε, θα μπορούσαμε να πάμε πιο μακριά, να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Ε, λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να σημειώσουμε ένα σημαντικό στοιχείο που υπόθηκε και νωρίτερα. Υπάρχει ανάγκη αποκατάστασης εμπιστοσύνης, να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των εργαζομένων και των περιφερειών, να νιώθουν ότι μπορούμε να τους βοηθήσουμε στην περίοδο αλλαγών, αλλαγών που τελικά είναι μόνιμες αλλαγές. Να μην υπάρχει προστατευτισμός και εθνικισμός σε αυτή τη συζήτηση. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να εφαρμόσουμε μία πιο στρατηγική προσέγγιση, πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση, με ένα πλαίσιο αναφοράς. Εγώ αποφεύγω τον όρο ε, κώδικας δεντολογίας, αλλά θα έλεγα ένα πλαίσιο αναφοράς, το οποίο θα προωθεί τις ε, βέλτιστες πρακτικές και θα φροντίζει να εφαρμόζονται αυτές. Και έτσι ξαναρχόμαστε στην ιδέα που υπάρχει σε τρία σημαντικά έγγραφα της Επιτροπής που είναι η βιομηχανική πολιτική, η, η ενιαία πράξη και το full skills job. Σε αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θα ξεκινήσει διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους φέτος ακόμα. Πάνω σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό για τις αναδιαρθρώσεις. Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος μαζί σας. Αυτή θα είναι μια δύσκολη υπόθεση. Γιατί πρόκειται ουσιαστικά για τα προβλήματα απασχόλησης που έχουμε στην αγορά εργασίας. Το θέμα των αλλαγών της μετάβασης έχει να κάνει με τους μισθούς, με τις ε, θέσεις απασχόλησης, πράγματα τα οποία για κάθε εργαζόμενο είναι ζωτική σημασία. Και εμείς προσπαθούμε να πετύχουμε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στο ότι πρέπει να διευκολύνουμε την προσαρμογή των επιχειρήσεων και συγχρόνως πρέπει να διευκολύνουμε και την ε, μετάβαση των εργαζομένων. Και πώς μπορούμε να συμφιλιώσουμε αυτά τα δύο στοιχεία. Σας το είπα, θα είναι δύσκολη η συζήτηση αυτή. Ο Επίτροπός μου είναι πεπισμένος για τη δυσκολία αυτή Πάντως κάθε στοιχείο που μπορεί να διευκολύνει αυτή τη συζήτηση είναι κάτι θετικό. Να προσθέσω κάτι, να διευκρινίσω κάτι γιατί πρόκειται για χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που χρησιμοποίησαμε γι' αυτό. Το ελεγκτικό συνέδριο κατέληξε σε θετικά συμπεράσματα, που σημαίνει ότι μπορώ να καθησυχάσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων του και μπορώ εδώ να ευχαριστήσω και την ΑΕΤΙΣΗ και την ILO για την βοήθειά τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Πρέπει και εγώ να πω εδώ ότι ακόμα και αν δεν ήμασταν πολύ άριθμοι σε αυτή την αίθουσα, να ξέρετε ότι δίνω μεγάλη σημασία στην ανταλλαγή απόψεων που είχαμε είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι λιγάκι το περιθώριο λιγμών που έχουμε. Ώστε να μην κάνουμε business as usual, αλλά να δούμε πού πρέπει να καινοτομήσουμε, προς τα πού πρέπει να πάμε, να είμαστε εμείς προδραστήριοι. Γιατί ξέρουμε ότι πρόκειται για μια δύσκολη δουλειά, ένα δύσκολο εγχείρημα και συχνά βλέπουμε ότι η απόσταση ανάμεσα στις προσδοκίες και την εφαρμογή είναι μεγάλη. Άκουσα αυτά που είπατε για την παρακολούθηση των συστάσεων από τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και το ΙΤΕ για την έρευνα αυτή, για τη δουλειά τους. Καλό θα ήταν βέβαια να έχουμε περισσότερους συναδέρφους εδώ κάθε φορά που ακούμε τα αποτελέσματα μιας πιλωτικής έρευνας. Για μας, που παίρνουμε την πρωτοβουλία, από κοινού βέβαια με την Εκτελεστική Επιτροπή, είναι σημαντικό να ξέρουμε τα αποτελέσματα μιας τέτοιας έρευνας πώς εφαρμόζονται στην πράξη. ιδίω όταν μιλάμε για βιομηχανική αναδιάρθρωση. Είναι πράγματα τα οποία εξακολουθούν να μας καίνε και με το οποίο θα έρθουμε αντιμέτωποι και τις επόμενες χρονιές. Σας ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά όλους και τους τρεις για τη συμμετοχή σας στην συνεδρίασή μας σήμερα το πρωί. Συνεπώς, εδώ κλείνει η συνεδρίασή μας για το πρωινό. Θα τα ξαναπούμε στις 3 μετά το μεσημέρι.